Good Καλημέρα. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, εγκρίνεται. Περνάμε σε ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Πρώτη ανακοίνωση. Αφορά τις ομάδες εργασίας για την οικονομική αρρωγή, αυτή την ομάδα εργασία, όπου αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εργασία που θα αποτελείται από 18 μέλη τη ΕΚΟΝ και 4 μέλη από άλλε επιτροπέ. 6 από το ΕΛΚΑ, 5 από του Σοσιαλιστέ, 3 από το ΡΙΝΙΟΥ, 2 από του Πράσινου, 2 από το ID, 2 από το ECR, 1 από την ΚΟΕ και 1 από του μη εγγεγραμμένου κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις άλλες ομάδες εργασίας. Ε, έλαβαν γνώση οι συντονιστές των ορισμών στις διάφορες ομάδες εργασίας. Τώρα για τις πολιτικές προτεραιότητες για την νέα θητεία και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αποφασίστηκε να ζητήσουμε την άδεια για διάφορες ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, τόσο νομοθετικές όσο και μη ε, νομοθετικές. Αποφασίστηκε ότι οι τίτλοι όμως και το περιεχόμενο θα προταθούν στην επόμενη συνάντηση επισκέψεις και αντιπροσωπείες της ΕΚΟΝ μέσα στο 2020. Η σύνθεση των ε, επισκέψεων στην Φραγκφούρτη και στην Βασιλεία αποφασίστηκαν τα εξή για τη Φραγκφούρτη. ΕΛΚ 3, σοσιαλιστές 3, δύο από το Ρινιού, ένας από τους Πράσινους, ένας από το ID, ένας από το ECR, ένας από την ΚΟΕ. Βασιλεία τρεις από το ΕΛΚ, τρεις από τους σοσιαλιστές, δύο από τη Ρινιού, ένας από τους πράσινους, ένας από τους ID, ένας ECR και ένας μη εγγεγραμμένος. Συμφωνήθηκε ότι στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ο κανόνας εκπεριτροπής DONT και στα διάφορα αποφασίστηκε να ζητήσουμε μια αλλαγή στον τίτλο της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για το εξάμεινο, αντί να λέγεται όπως τώρα Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την, ε, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, να είναι Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2020. Έχω κρυώσει, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Τρίτο σημείο. Έκθεση για τι ε, συνεχιζόμενε διοργανικέ διαπραγματεύσει όσον αφορά του φακέλου για τη συμμετοχική χρηματοδότηση. Στι 18 Δεκεμβρίου του 2019 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά δύο νομοθετικά κείμενα για το θέμα αυτό. Συνεχίζεται τεχνική ε, εργασία και θα ψηφίσουμε αργότερα. Η προσωρινή συμφωνία βασίζεται στο αποτέλεσμα πέντε τριμερών διαλόγων με βάση τα κείμενα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αναθεωρήθηκαν από την ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Διάφορα θέματα στο οποία δεν έχουμε συμφωνήσει έχουν να κάνουν με το όριο της σημαντικής ε, χρηματοδότησης, με την προστασία των επενδυτών, με τα χρονικά όρια και το ρόλο της ΕΣΜΑ. Άλλο θέμα οι βιώσιμες επενδύσεις. Είναι θέμα που εξετάζουν από κοινού η ΕΚΟΝ και η Στο 16 Δεκεμβρίου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξε προσωρινή συμφωνία για το σύνολο του νομοθετικού κειμένου. Η ΕΚΟΝ και η ΕΝΒΙ θα ψηφίσουν από κοινού αύριο μετά από την ε, διαδικασία ε, δεύτερης ανάγνωσης. Η προσωρινή συμφωνία βασίζεται στους τριμμένους διαλόγους 3 και 5 Δεκεμβρίου και οι διαπραγματευτικές ομάδες κατέληξαν σε συμβασμούς για θέματα κλειδί, όπως έχουν να κάνουν τις εγκάρσιες δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις ε, δημοσιοποίησης, την δημιουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση την ε, χρήση των κατεξοδότηση πράξεων, ε, τον αποκλεισμό των ε, ορυκτών καυσίμων κτλ. Στις 16 Δεκεμβρίου επιπλέον θέματα διευκρινίστηκαν και συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο βάσει του άρθρου 12 που καθορίζει πώς οι οικονομικές δραστηριότητε μπορούν να βλάψουν τους στόχους μας για το περιβάλλον. Το επόμενο θέμα είναι έγκριση των πρακτικών. Πρακτικά της 18 Δεκεμβρίου 2019 ε, Δευτέρας και 3 Δεκεμβρίου 2019 και 12 Δεκεμβρίου 2019. Ε, συνεχίζουμε, περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι Ευρωπαϊκό Εξάμενο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2020. Η εισηγήτρια είναι ο Ρόρ Λαλούκ από τους σοσιαλιστές. Και μετά έχουμε τους κοιόδης ογητές, Γκιόρη από το ΕΛΚ, Έρογλου από το Ρινιού, Λάμπερτς από τους Πράσινους, Γκούντερ Μπέκ ID και Τσίκα ECR. Έχουμε συνδεδεμένη επιτροπή, την Επιτροπή Προπλογισμών και γνωμοδοτήσει από την Ένβη, Ρέγγι και Γυναίκες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λαλουκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Ε, καλή ανάρρωση καταρχήν και ε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις του περιβάλλοντος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις ε, νομιμοποιούμενες, νόμιμες ε, αγωνίες των Ευρωπαίων πολιτών και ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μας, αλλά και πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, ε, ο ΑΣΕΜΑ ζητούν να αδράσουμε. Και πριν από το Νταβός ε, κατάταξαν τις πέντε βασικές γεωπεριβαντολογικές ε, αγωνίες που είναι η απώλεια της βιοπικιλότητας, οι φυσικές καταστροφές, τα μετεωρολογικά φαινόμενα που είναι βία, όπως επίσης και η δυνατότητα των δημοσίων φορέων να αντιμετωπίσουν ε, ταχύτατα και με αποτελεσματικότητα αυτά τα φαινόμενα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στον Ταβός και είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε ε, να αντιδράσουμε σωστά και γρήγορα. Είναι ε, πολύ σημαντική αυτή η απειλή, είναι σοβαρή και μέσω της ε, Προέδρου του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος, η Ευρώπη, μέσω της δυνατότητας μετάβασης σε ε, ε, μια κλιματικά θετική πολιτική με μια στεναρή φωνή ε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί στο ευρωπαϊκό εξάμεινο να εντάξουμε κάποιες πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να συμμορφωθούμε με αυτό το στόχο. Έτσι ώστε θα πρέπει οι πολιτικές μας να λαμβάνουν υπόψη την πτυχή την κοινωνική και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα κριτήρια της έκθεσης και μέσω της έκθεσης εμείς θέλουμε να υπογραμμίζουμε πως στηρίζουμε και πλαισιώνουμε το ε, Green Deal ότι το εξάμεινο λαμβάνει υπόψη στόχους περιβαλλοντος αλλά και οικονομικού, γιατί το περιβάλλον έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία και επίση ε, να έχουμε ε, συνέπεια με τον τίτλο τον οποίο δώσαμε σε αυτό το εξάμεινο και στην έκθεσή μα που θα είναι η ανάπτυξη, ε, η βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συντονίσουμε όλες τις οικονομικές πολιτικές με έναν τρόπο έτσι ώστε να έχουμε μια μετάβαση κοινωνική, οικολογική, με ε, για το περιβάλλον, για την ε, ευημερία, για την μάχη κατά της ένδυας τη κοινωνική οικονομική αλλά και τη περιβαλλοντολογική, να δούμε τι θα γίνει με τα αέρια του θερμοκηπίου και πώς μπορούν να περιοριστούν, να εντάξουμε σε αυτό και στις οικονομίες μας στην παγκόσμια οικονομία και να δούμε τι θα γίνει ε, με τα επίπεδα εκπομπών τα οποία επίση προσπαθούμε να μετριάσουμε. Επίσης, έχουμε την ε, βούληση να επιλέξουμε και ένα χρυσό κανόνα για τις επενδύσεις, γιατί πια η κρίση του περιβάλλοντος είναι ε, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να πιστέψουμε πω διακυβεύεται η ίδια η επιβίωσή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να ισχύει και στις ιδιωτικέ επενδύσει με στα κράτη-μέλη. Η ζώνη του ευρώ εδώ και χρόνια πλήττεται από υποεπενδύσεις ε, στις ε, διαστοτικές δράσεις, κάτι το οποίο ε, επισημαίνουμε σε κάθε έκθεση για το εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν οι συλλογικέ υποδομές, η παιδεία, η επιστήμη και η έρευνα, όπως μας λέει και όσα, να λάβουν υπόψη οικονομικές πολιτικές που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, αλλά θα επιτρέψουν και οικονομίες μας να προσαρμοστούν στις προκλήσεις τούτου του αιώνα. Αν λοιπόν ε, ε, οι επιδόσεις μας βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, παράλληλα διαπιστώνεται και μια αύξηση της ανισότητας, περισσότεροι ε, εργαζόμενοι που ζουν ε, στη φτώχεια και χειροτέρευση της ποιότητας ζωής. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη της οικονομίας δεν συνεισφέρει επαρκώς στην βελτίωση της κοινωνικής, ε, του κοινωνικού περιβάλλοντος στη ζώνη του ευρώ. Και οι πολιτικές που μέχρι στιγμής έχουμε λάβει ήταν φιλόδοξες και είχαν στόχο και φιλοδοξία να αναζωπυρώσουν τις οικονομίες μας και να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν το πέτυχαν. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέσω του ε, Green Pact. Θέλουμε να αναμορφωθεί και η τραπεζική νομοθεσία έτσι ώστε να έχουμε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για να έχουμε ένα περιβάλλον οικονομικό σταθερό που θα βασίζεται στον υγιή και όχι στον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Έναν ανταγωνισμό ο οποίος δεν θα αφήσει ε, και θα στερήσει από τα κράτη και από τους πληθυσμούς πόρους οι οποίοι είναι κρίσιμη για τη μετάβαση σε, μια καλύτερα οικολογική, ε, σε ένα καλύτερο οικολογικό ε, περιβάλλον οικονομικό. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, όλοι εμείς θα πρέπει να ε, λάβουμε μέρος στο διάλογο αυτό και γι' αυτό εμείς επιμένουμε στην ανασωπήρωση του διαλόγου που θα λαμβάνουν μέρος και η ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πλήρως πώς το περιβάλλον είναι ένα θέμα που επήγε. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές της έκθεσης. Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσω να συνεργάζομαι με τους κοιόδης. Ξέρω πως οι συζητήσει θα είναι ενθουσιώδεις, θα είναι πλούσιες, θα είναι γεμάτες. Και ένα κοινοβούλιο το οποίο θέλει να έχει βορνή θα πρέπει ε, να ε, δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το θέμα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε τώρα το λόγο στους Σκιώδης. Νίκο από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά μαζί πιστεύω. Μέχρι ότου να λάβει την τελική της μορφή αυτή η έκθεση είναι σημαντική η προσπάθεια. Το 2011 Τότε εγώ ήμουν υπουργό ε, για ευρωπαϊκά θέματα κατά την Ουγγρική ε, Προεδρία. Τότε έζησα το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, οπότε έχω μνήμες από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι το εξάμεινο θα πρέπει να διατηρηθεί ως ολοκληρωμένο εργαλείο για τις οικονομικές ε, πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης. Δίνει κατεύθυνση στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες Έχουμε αποκλειστικέ αρμοδιότητε κρατών μελών, σύνθετε αρμοδιότητε και ευρωπαϊκέ αρμοδιότητε. Οπότε όταν δίνουμε κατεύθυνση και οδηγίε, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Φυσικά, εκτιμώ το ότι η συγγήτρια θέλει να προσαρμόσει την έκθεση ε, στα νέα κατεπήγοντα θέματα, στο κλίμα, στην πράσινη συμφωνία, τα οποία έχουν υψηλή προτεραιότητα το κοινοβούλιο μας κάθε μήνα υιοθετεί τουλάχιστον μία έκθεση για τα θέματα αυτά, παρότι δεν λένε πάντα το ίδιο πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι για να αλλάξουμε πλήρω την εστίαση και να βάλουμε στο επίκεντρο την Πράσινη Συμφωνία, υπάρχει κίνδυνο ε, να επαναλαμβανόμαστε σε διάφορε εκθέσει και να χάσουμε την ουσία τη παρουσία εκθέσης. Οπότε η σύστασή μου θα ήταν να διατηρήσουμε τον αρχικό σκοπό του Ευρωπαϊκού Εξαμένου που όπως είπα ήταν να παρέχει κατεύθυνση για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, υπάρχει μια πρόταση που πιστεύω ότι υπάρχει σε πολλές ε, γλώσσες ε, ότι όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Οπότε θα λέτε ότι πρέπει να εστιαστούμε στην Πρασινή Συμφωνία, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την εξορρόψη των φύλων. Δεν βλέπω να είναι εξισορροπημένη όλη αυτή η αντιμετώπιση. Άρα σκεφτούμε τι έχει ήδη υιοθετηθεί και το τι έχει συμφωνηθεί αρχικά. Μια άλλη σκέψη δική μου προς την εισηγήτρια. Φυσικά θα λάβουμε γνωμοδότηση από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης την οποία θα πρέπει να προσαρτήσουμε στην εκθεσή μας και να εντάξουμε και τις δικές τους ε, συστάσεις και παρατηρήσεις. Στην εκθέση αυτή λοιπόν εγώ θα έλεγα να εστιαστούμε περισσότερο στις δικές μας αρμοδιότητες ως επιτροπή ΕΚΟΝ. Μια άλλη σκέψη είναι ε, η οικειοποίηση. Αναφέρατε κι εσείς ε, η συγγήτρια πόσο σημαντική είναι η οικειοποίηση γιατί αν τα κράτη-μέλη δεν θεωρούν ότι είναι δικό τους το θέμα Απλά θα το σημειώσουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Ο στόχος του να κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό ε, είναι να το λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη. Όπως ε, είπα και προηγουμένως, αν χάσουμε την εστίαση θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά αυτή την οικειοποίηση. Μας περιμένουν δύσκολες συζητήσεις ε, για τον κανόνα, για τα σύνορα, για τα συστήματα απασχόλησης που δεν είναι νέα ζητήματα και δεν πιστεύω ότι θα επιληθούν μέσα από αυτή την έκθεση. Οπότε επαναλαμβάνω ως βασική μου παρατήρηση να επικεντρωθούμε στα βασικά ζητήματα. Και έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή βιώσιμη έκθεση την οποία θα λάβουν και υπόψη τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγγενερόγλου από το Ρινιού. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Λαλούκ, σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση. Όταν τη διαβάζει κανείς, έχετε εργαστεί εντατικά, διότι βλέπει κανείς ότι τελικά το πνεύμα και η αιστείες αυτής της έκθεσης έχουν αλλάξει τελείως. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολλές ώρες που σίγουρα περάσατε και επενδύσατε για αυτή την έκθεση. Ε, δυστυχώς όμως ε, βλέπουμε ότι έχετε αλλάξει το πνεύμα της έκθεσης. Και η έκθεση η οποία αρχικά αφορούσε ε, το να, δίνουμε, να αφήνουμε τον έλεγχο στα κράτη-μέλη έχει αναδιατυπωθεί και είναι ένα έγγραφο αιτήσεων ουσιαστικά σε αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές άλλες εκθέσεις. Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε, αλλά σε τελική ανάλυση ε, δεν είναι το θέμα αυτής της έκθεσης. Δηλαδή κάνατε πολύ καλή δουλειά, αλλά σε λάθος έκθεση. Εμείς ως Ρενιού θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποβάλουμε ε, τροπολογίες ώστε να επιστρέψει η έκθεση στο παλιό της πνεύμα. Να μην χτίζουμε ιδεολογικούς ε, τείχους αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν θέλουν να γίνει μια πράσινη συμφωνία. Δεν χρειάζεται ε, ένα τέτοιο έγγραφο. Ε, ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό έτσι και σα απευθύνω έκκληση. Ε, αφήστε να γίνει η Πράσινη Συμφωνία σε άλλε εκθέσει, όχι σε αυτήν εδώ. Όσο και αν είναι αξιόλογη η εργασία σας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να βρούμε μια καλή ε, συμβιβαστική λύση. Ε, εμείς λάβαμε την εκθέση στις 16 Ιανουαρίου τώρα για τα διαδικαστικά και δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες ε, ψηφιακά, πρέπει να τις στείλουμε όλες γραπτά. Αυτό είναι πάρα πολύ δουλειά ε, και με τη διοίκηση. Οπότε στρέφουμε τώρα και στην ε, Πρόεδρο. Θα έπρεπε να μπορούμε να υποβάλουμε ψηφιακά τις, ε, ηλεκτρονικά τις ε, τροπολογίες όπως κάνουμε και σε άλλες ε, εκθέσεις. Αλλιώς είναι πάρα πάρα πολύ δουλειά το να πρέπει να τα γράψουμε με το χέρι και να τα υπογράφουμε με το χέρι. Υπάρχει ο ψηφιακό τρόπο και ελπίζω η κυρία Λαλούκ να μπορέσει να συμφωνήσει. Ευχαριστώ πολύ. Για να μπορέσουν να ενταχθούν και οι δικέ μα απόψει μέσα σε αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Φιλίπ. Λαμπέρτ τώρα από τους πράσινους. Όταν δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια το εξάμεινο, το υποστηρίζαμε πολύ, γιατί πιστεύαμε ότι έτσι θα συντονιζόταν καλύτερη οικονομική πολιτική και είναι σωστό να πούμε ότι πολλές ε, πτικές οικονομικής και κοινωνικής ε, πολιτικής ε, συντονίζονται καλύτερα που ήταν αρμοδιά των χωρών μελών η επιμερισμένη ευθύνη. Δεν είναι όπως στη Σοβιετική Ένωση που από πάνω καθορίζονται τα πράγματα. Για χρόνια όμως η υπόθεση που κάναμε για το εξάμενο είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες δεν ξεπερνάν τα όρια, κάτι το οποίο είναι μια απειλή για μια εύρωστη οικονομία. Και αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει, πρώτα απ' όλα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, και δεύτερον ότι τι νόημα έχει να έχουμε μια οικονομία αν αυτή δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Και θυμάμαι ότι ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚΑ ε, ήταν υπεύθυνο για την οικονομία που εξυπηρετεί το κόσμο, αλλά ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Περισσότεροι το καταλαβαίνουν αυτό. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και το εξάμεινο αποτελεί μία δοκιμή για να χρησιμοποιήσουμε τελικά την τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία. Γιατί πρόκειται για συμβιβασμούς και τελικά η έκθεση γίνεται ε, χωρίς, έτσι γινόταν στο παρελθόν τουλάχιστον, χωρίς ε, ανάμειξη ανθρώπων. Βάσει των αριθμών καταλήγαμε στα συμπεράσματα. Τώρα έχουμε την Πράσινη Συμφωνία. Που είναι φιλελεύθερη, δεν ξέρω, α, ναι, δεν ξέρω το όνομά σας ακόμα, αλλά το είπε ότι δεν είναι σαν έχουμε ένα κουτάκι που λέγεται πράσινη συμφωνία και το κρατάμε απομονωμένο από τις υπόλοιπες πολιτικές μας. Όχι, να είμαστε σοβαροί. Η πράσινη συμφωνία τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνίες έχουν μέλλον και για να έχουν μέλλον πρέπει να σεβαστούμε ε, τα όρια που μας βάζει ο ίδιος ο πλανήτης και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέσα σε αυτά τα ε, όρια μπορεί να, να ζήσουν όλοι. Οπότε συμφωνώ με την εισηγήτρια. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αν το εξάμενο το αποσυνδέσουμε από αυτό, ε, λειτουργούμε σχιζοφρενικά και πρέπει να το αντιληφθούμε. Και οι δικές μας τροπολογίες θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε συνεπείς πολιτικές. Το, η νέα πράσινη συμφωνία δεν είναι κάτι μοδάτο, κάτι που πρέπει να το λέμε, όχι. Είναι για να κατευθύνει τις πολιτικές μας. Και πάλι, και επιμένω πάνω σε αυτό, ε, κοιτώντας και τους συναδέρφους του ΕΛΚΑ, να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες των χωρών μελών, των περιφερειών, γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα. Αν προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε, ε, αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για να αποτύχουμε. Πρέπει να χτίσουμε συγκλήσεις και συμφωνίες. Και πράγματι, όλοι πρέπει να συμφωνήσουν για το ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να υλοποιηθεί και τα προβλήματα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στις χώρες μέλη, στις περιφέρειες. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί αυτός ο ενθουσιασμός που θα οδηγήσει στις συγκλήσεις. Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα και αυτό είναι το δικό μας πνεύμα των πρασίνων. Πρέπει να αρχίσουμε να επανακατευθύνουμε τις πολιτικές. Όχι να λέμε ότι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα ήταν σαν όχι. Αλλά αν μη τι άλλο να αναγνωρίσουμε τα όρια των πολιτικών που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε βγει από τι δυσκολίες. Και για αυτούς που πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση, ε, να ξέρετε ότι σήμερα είμαστε σε χειρότερα επίπεδα από ό,τι είμαστε πριν από την ε, ε, η οικονομική κρίση. Και εδώ πέρα πρόκειται για το ιδιωτικό χρέος. Δείτε τα δάνεια των ε, φοιτητών, ε, των εταιριών. Όλα αυτά τα δάνεια δεν πρόκειται να αποπληρωθούν. Κάποια δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Οπότε για σας που πιστεύετε ότι υπάρχουν μόνο κάποιοι ανεύθυνοι και εδώ στρέφω προς τους φιλελεύθερους και ότι αυτοί οι ανεύθυνοι είναι τα κράτη, όχι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλοί που συμπεριφέρονται ανεύθυνα. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική που λέει ότι τα κράτη φταίνε, αυτή είναι κακή. Να δίνουμε την ευθύνη πραγματικά εκεί που αναλογεί, όσο αναλογεί στον καθένα. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω τον κύριο Πεκ από το ID. Υπάρχει κάποιος άλλος μήπως που θέλει το λόγο. Όχι. Ωραία. Α, παρακαλώ. Εσεί ναι. Φρανσίσκα Ντονάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμένα μου αρέσει πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την έκθεση στην ε, εισηγήτρια την κυρία Λαλούκ. Πιστεύω ότι έχει ασχοληθεί με τα βασικότερα θέματα το περιεχόμενο αυτής της πρότασης ε, τραβά την προσοχή στα βασικά σημεία ώστε να αλλάξει μορφή η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της ε, μακροοικονομικής ισορροπίας με μια νέα προσέγγιση η οποία σε τελική ανάλυση λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, την ανάγκη αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη και να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο, δίνοντας περισσότερη προσοχή στο ιδιωτικό χρέο, όπως είπε ο συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα πολύ σωστά, σε σύγκριση με το δημόσιο χρέο που εξετάζουμε μόνο μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν συγχαρητήρια στη συνάδελφο και είμαι βέβαιη ότι η προσπάθειες που θα ακολουθήσουν και η δουλειά, που θα γίνει με τις τροπολογίες θα οδηγήσουν σε μια έκθεση υψηλής ποιότητας που θα τύχει ευρεία συμφωνία. Σε ευχαριστούμε. από το ECR παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Αντιλαμβάνομαι αυτά που τονίζει και την αποφασιστικότητά της για τα πράσινα ζητήματα και την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Είναι σημαντικά θέματα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη ισορροπία στην έκθεση αυτή, ώστε να δώσουμε σημασία και στα σημερινά προβλήματα των ευρωπαϊκών οικονομιών, που μπορεί να επιδεινωθούν στο μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε τρία ζητήματα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, επενδύσεις. Ναι, το επίπεδο επενδύσεων είναι κάτω από τα επίπεδα που είχαμε πριν από την κρίση. Και ναι, χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε κάποιους τομείς, περισσότερο από άλλους, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ακριβώς κάποιες επενδύσεις είναι που οδήγησαν τελικά στην τελευταία κρίση. Το θέμα είναι η αξία του χρήματος που παίζει σημαντικό ρόλο και όχι η ενώ ονομαστική τους αξία. Οπότε διαφωνώ για το ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και ότι αυτό πρέπει να αποτελεί άλοθη για περισσότερη ευελιξία τελικά ε, όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, γιατί αυτό τελικά θα οδηγήσει σε περισσότερο δημόσιο χρέος κατά πάσα πιθανότητα, κάτι το οποίο έτσι κι ήδη βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα που είχαμε πριν από την κρίση. Έπειτα να προσέξουμε περισσότερο και το θέμα της ε, μεγέθυνσης, της ανάπτυξης. Βλέπουμε τα επίπεδα ανάκαμψης και τι θα περιμέναμε μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης. Αλλά χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας δεν πρόκειται να λύσουμε τα θέματα της βιωσιμότητας ή των ε, δημοσίων οικονομικών στις χώρες μέλη. Λαμβάνοντας κυρίως υπόψη και το δημογραφικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολιτικές που οδηγούν σε μηδέν ε, επιτόκια, να τα ξεχάσουμε και να φτάσουμε σε κανονικά επίπεδα επιτοκίων όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί μόνο έτσι θα αναγκαστούν και οι χώρες να εφαρμόσουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Ε, κατά τα άλλα έχω επιφυλάξει για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε φορολογικά ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει να κάνει με την έκθεση αυτή, όπως επίσης και κάποια άλλα. Για να μείνουμε ανταγωνιστικοί, οι χώρες μέλη πρέπει, για να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον έξω κόσμο, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και μεταξύ μας οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό μπορεί να γίνει, να έχουμε συγκρίσιμους ε, δείκτες ε, στα φορολογικά και πρακτικές. Και αυτός θα ήταν καλύτερος τρόπος προκειμένου τα φορολογικά μας συστήματα να είναι πιο ανταγωνιστικά. Θα περιοριστώ σε αυτά τα σημεία. Ίσως να μην ευχαριστώ με τις απόψεις μου την εισηγήτρια, αλλά προσβλέπω σε επικοδομητικές συζητήσεις σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Μη γκούε τώρα. Παρακαλώ, κύριε Κουσμάου. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συζητήσει πάρα πολύ συχνά το θέμα της ε, ανάπτυξης που αναμένεται. Το πράσινο πακέτο έχει παρουσιάσει νέες κοινωνικές πολιτικές, έχει στόχους για το περιβάλλον που είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, αλλά δεν έχουμε νέους ε, χρηματοδοτικούς πόρους για να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς με ποιο τρόπο θα πετύχουμε όλους αυτούς τους νέους στόχους που έχουμε θεσπίσει. Και βέβαια εδώ έχουμε και ένα στόχο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά ε, σωστός, που είναι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, γιατί είδαμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι, πώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά χωρίς τους πόρους που μας επιτρέπουν να πετύχουμε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε. Χρειαζόμαστε επένδυσεις, επενδύσεις σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή επενδύσεις και από τα κράτη-μέλη. Αν όλοι αυτοί οι στόχοι, τους οποίους επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, αύξηση μισθολογική, κάτι το οποίο τελευταία δεν διαπιστώνουμε να ε, σημειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν λοιπόν όλοι αυτοί οι στόχοι δεν εμφανίζονται στις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τότε οι προσπάθειες αυτές είναι κενές, στερούνται νοήματος και επίσης κενή είναι και οι στόχοι τους οποίους περιγράφουμε. Δηλαδή, Στη συζήτηση που κάνουμε για την έκθεση αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες, δεδομένου ότι δεν έχουμε επιπρόσθετους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τους πετύχουμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για τα κομμάτια που ανήκουν στο χώρο της συνοχής, εδώ οι πόροι θα μειωθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει η εθνική πολιτική να δώσει την απάντηση και θα σας εξηγήσω τι γίνεται στη δική μου χώρα. Τα τελευταία χρόνια μειώσαμε με ε, τρόπο άνευ προηγουμένου το δημόσιο χρέος και πώς το κάναμε, όχι μέσω λιτότητας, αλλά μέσω αναπτυξιακών πολιτικών. Και θα ήθελα να απευθύνω και μια δεύτερη ερώτηση, η οποία σχετίζεται με ένα θέμα το οποίο δεν περιγράφεται καλά στην έκθεση, η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται σχεδόν πάντα στις συγκεκριμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν είναι και πια τόσο συγκεκριμένες. Δηλαδή η κατάργηση των ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εκεί, όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να μάθουμε αυτή η κατάργηση των ρυθμίσεων. Τι έφερε ας πούμε στους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποιο ήταν ο αντίκτυπος που είχε. Επίσης, Οι εργασιακές σχέσεις είναι ε, ε, πλέον σε εξαιρετικά δεινή θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κινδυνεύουν να καταστραφούν. Θέλω τώρα να στραφώ και στα, στις μακροοικονομικές ε, ανισότητες και στην έλλειψη ισορροπίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελούν τεράστια πρόκληση άνευ και που αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μάλλον γραφειοκρατικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται και αυξάνονται οι επενδύσεις όταν οι χώρες έχουν πλεονάσματα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν έχει ε, αλλάξει γιατί οι χώρες οι οποίες έχουν πλεονάσματα δεν αλλάζουν πολιτική αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοια εξωτερικά μεγάλα πλονέσματα για κάποιους όταν βρισκόμαστε σε μια οικονομική και νομισματική ένωση και έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι πάντα πλονισματικοί και κάποιοι οι οποίοι έχουν μονίμως ελλείμματα, πού είναι οι μεταβιβάσεις, Πού είναι τα εργαλεία τα θα, θα μας επιτρέψουν να εξομαλύνουμε την κατάσταση και να βοηθήσουμε. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει ε, με τα σχόλιά της το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες που διαβάσατε την έκθεση και που κάνατε κάποια πρώτα σχόλια. Ε, όντως, με τις τροπολογίες που λάβαμε ίσως θα καθυστερήσουμε κάπως, κυρίως για την οργάνωση της πρώτης ε, συνάντησης. Αυτό είναι το πρώτο βασικό τεχνικό θέμα που πρέπει να θέσω. Άκουσα ε, σχόλια, ε, έχω, άκουσα ορολογία για ισότητα, για ελλείμματα, για γυναίκες για μακροοικονομικούς στόχους, για εσωτερική ε, έλλειψη ισορροπίας, στοιχεία δηλαδή στα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε. Τώρα για το ποιο είναι το πνεύμα που διέπει το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ποιε είναι οι αρμοδιότητες και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου, γιατί καταλαβαίνω τον πειρασμό του να παραμείνουμε στο παλαιό πνεύμα του εξαμήνου και να τα κάνουμε όλα όπως τα κάναμε ε, στο παρελθόν με παραδοχές μακροοικονομικές και σενάρια, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει. Το περιβάλλον θέτει νέες προκλήσεις η οικονομία ε, δεν είναι μια βιοσφαίρα η οποία μας επιτρέπει, βιόσφαιρα με μας επιτρέπει να επιβιώνουμε έτσι εύκολα. Υπάρχει το θέμα του περιβάλλοντος και έχουμε και την απώλεια της βιοπικιλότητας. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εκτός, γι' αυτό χρειαζόμαστε τους δείκτες για το περιβάλλον ε, μέσα σε αυτό το κείμενο και θα βάλουμε ε, προτεραιότητες οι δείκτε οι οποίοι ανήκουν στη δική μου πολιτική ομάδα, του σοσιαλδημοκράτε, ίσως και κάποια φιλελεύθερου δείκτε, αλλά αυτή τη στιγμή ε, εξελίσσεται το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και μέσα στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να τεθούν κάποια θέματα σαν αυτά τα οποία προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είμαστε επραγματιστές και να μην πέσουμε σε ε, ιδεολογικές ε, αναζητήσεις. Είδα τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, βλέπω τις γενικότερες γραμμές που διαγράφονται, δηλαδή ε, ο χρυσός κανόνας, ε, θα συζητηθεί πολύ. Νομίζω ότι <laughs> βιάζομαι να ξεκινήσω για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το εξάμεινο για να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Νομίζω αυτό στόχο έχει η έκθεση που θα ε, συντάξω. Ευχαριστώ. Για να κλείσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι δεδομένης της προθεσμίας για τη διαδικασία πρέπει να ενημερώσω όλα τα μέλη ότι στις 16 Ιανουαρίου προβλέπεται, ε, αναβάλλεται η ημερομηνία ε, για προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 24 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια η έκθεση και στην ΕΚΟΝ πριν το ΕΑΡΙΝΟ Συμβούλιο. Δηλαδή θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ε, η ηλεκτρονική υποβολή τροπολογιών δεν είναι δυνατή διότι η ΕΚΟΝ ε, απαιτεί να υπάρχουν όλες οι μεταφράσεις και επειδή 9 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε η έκθεση μεταφράσεις δεν θα είναι έτοιμες πριν από τις 24 Ιανουαρίου που είναι και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Γι' αυτό υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα, λυπάμαι, αλλά η διαδικασία αυτή τη φορά είναι αυτή. Το επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη είναι στι 10, οπότε θα πρότεινα να κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, που είναι οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Στράφκο Μαρίτς, που είναι ο πρόεδρος της ε, ΕΚΟΦΗΝ και αναπληρωτής ε, πρωθυπουργός της ε, Κροατίας και υπουργός οικονομικών. Έχει αναλάβει την εκπεριτροπής προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ από 1η Ιανουαρίου και δέχτηκε να έρθει και να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας σε θέματα της Επιτροπής μας. Η Προεδρία της Κροατίας λαμβάνει χώρα σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή, τώρα που έχουμε και τη νέα Επιτροπή. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Κροατική Προεδρία για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Οπότε, σύμφωνα με την πρακτική μας, θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, εισαγωγικέ παρατηρήσεις από τον κύριο Μάριτς για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια 5 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις με τη δυνατότητα επερώτησης εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος στο διάστημα που προβλέπετε. Στον πρώτο γύρο ε, οι πολιτικές ομάδες και μετά θα ακολουθήσουμε με το σύστημα DON'T για τη σειρά των ερωτήσεων από τι πολιτικές ομάδες. Και αν μα το επιτρέπει ο χρόνος, θα υπάρξουν επιπλέον ερωτήσεις σε διαδικασία Catch Παρακαλώ κύριε Μάριτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Σινιάλη. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ, κύριε και κύριοι, βρίσκομαι εδώ με πολύ χαρά και είναι και τιμή μου εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της κρατικής προεδρίας στον τομέα των ε, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων. Η Κροατία αναλαμβάνει την προεδρία ε, σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Το γενικό περιβάλλον είναι περίπλοκο και απρόβλεπτο. Υπάρχουν επιπλέον προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, του μεταναστευτικού, του δημογραφικού, των παραπληροφοριών που κυκλοφορούν, του ανερχόμενου λαϊκισμού, τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός αυτής. Επίσης αντιμετωπίζουμε προκλήσεις εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον οικονομικό χώρο σαφώς και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα επίπεδα τα χαμηλά ανάπτυξης και οικονομικές διαφορές. Αυτές είναι κάποιες ανησυχίες που πολύ σωστά οι πολίτες μας περιμένουν από μας να αντιμετωπίσουμε. Επιπλέον, βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου θεσμικού και νομοθετικού κύκλου, κάτι το οποίο προσφέρει νέες Ευκαιρίε για να ξαναδούμε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανανεωμένη ενέργεια. Η Κροατική Προεδρία είναι έτοιμη από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει προς τους στόχους αυτούς. Τώρα θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποιες παρατηρήσεις για την οικονομική κατάσταση. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επέκταση που ξεκίνησε το 2013 συνεχίζεται, παρόλο που η μεγένθηση επιβραδύνεται ιδιαίτερα από το 2018 και μετά. Συγχρόνως υπάρχουν κάποια ε, μηνύματα που μας στάνουν για κάποια σταθεροποίηση στην καθοδική αυτή πορεία. Η τελευταία πρόβλεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει το Ευρωπαϊκό ΑΕΠ να αυξάνει κατά 1,4% το 2020 και 2021, κάτι το οποίο δεν αλλάζει από το 2019. Οι κίνδυνοι όμως που ελοχεύουν όσον αφορά την σπροπτικές μεγένθησης ε, παραμένει σε καθοδική πορεία. Ε, το καλό νέο είναι ότι δεν είναι τόσο έντονη η κίνδυνη αυτή. Έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε την ύφεση, αλλά είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι λιγότερο έντονοι, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί. Συνεπώς, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε και να συντονίσουμε την δράση μα αν αυτή η επιβράδυνση επιδεινωθεί. Πρέπει να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να τις κάνουμε περισσότερο ανθεκτικές και να είναι έτοιμες σε τριγμούς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης των οικονομιών μας, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, κάτι το οποίο απαιτεί προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, επ' αυτού, η τόσα μας ε, έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2020 είναι πολύ σημαντικά. Μαζί με την Προεδρία του Eurogroup θα οργανώσουμε σε βάθος εξέταση των συστάσεων στην Ευρωζώνη και θα ζητήσουμε την έξι του Συμβουλίου. Επίσης θα προχωρήσουμε και με τις αναχώρα συστάσεις για όλες τις χώρες ε, μέλη. Προβλέπουμε επίσης στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία που αφορά τα λεγόμενα το πακέτο των δύο και των 6 οδηγιών. Είναι αναγκαίο πολύ γρήγορα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο που θα κατευθύνει τις εθνικές μας και ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαι σίγουρος ότι η έκθεση αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα για σε βάθος συζητήσεις τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα δώσουμε και συνέχεια ανάλογα με τα συμπεράσματα. Τώρα, η εφαρμογή των συστάσεων και ο συντονισμό βάσει κανόνων των εθνικών πολιτικών είναι ζωτική σημασία. Αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι τη ιστορία αυτό, γιατί πρέπει να προδεύσουμε και όσον αφορά την εμβάθυνση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση και των ε, βασικών τη στοιχείων. Εμεί, ω Προεδρία του Συμβουλίου, έχουμε δεσμευτεί πέρα αυτού. Και δεν πρόκειται μόνο επειδή η Κροατία σκοπεύει να ακολουθήσει το ευρώ, να έχει το ευρώ σε λίγα χρόνια, ξέρετε ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει με τον στόχο αυτό να έχουμε το ευρώ, αλλά και επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι μια καλώ λειτουργούσα οικονομική και νομισματική ένωση είναι προ το συμφέρον όλων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε στενά επίσης με το Eurogroup, που έχει εντολή από του ηγέτε μα να ακολουθήσουν επίσης αυτή την πορεία και να την προωθήσουν. Θέλουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα αναθεώρησης και επενδύσεων που αποτελεί και τον προπολογισμό βασικά για την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη. Επίσης και το μέσο για την σύγκληση και την μεταρρύθμιση για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης και την τεχνική αρρωγή. Το νομοθετικό έργο επίση συνεχίζεται και παρακολουθούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ε, επίσης και τον προπολογισμό για την ε, σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα που συμφωνήθηκε στο Eurogroup τον Οκτώβριο μας πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό να ε, προχωρήσουμε και είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν βάλει από κοινού την κυριαρχία τους όσον αφορά την νομισματική πολιτική και τον μηχανισμό ισοτιμιών. Σίγουρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον τριμερή μας διάλογο, να τον ξεκινήσουμε μάλλον, για την μεταρρύθμιση και την στήριξη στις επενδύσεις ήδη αυτό το εξάμεινο. Τώρα ένας άλλος τομέας που μας απασχολεί είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Στόχος μας πρέπει να είναι σταδιακά να προχωρήσουμε προς τον τραπεζικό τομέα με καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων, με λιγότερους κινδύνους, με περισσότερο επιμερισμό κινδύνων και να συμπεριλάβουμε σε όλα αυτά και το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων. Η πρόοδο όσον αφορά το τελευταίο το έντις δεν έχει προχωρήσει πολύ. Αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να το κάνουμε και να ξεφύγουμε από τα διέξοδα. Οποιαδήποτε πρόοδο στο θέμα αυτό απαιτεί συζητήσεις σε βάθος και για χρόνο. Εμείς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές σε συνεργασία με την Προεδρία του Eurogroup. Ένα άλλο βασικό θέμα που μας απασχολεί για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι να αντιμετωπίσουμε και την κληρονομιά που μας άφησε η πρόσφατη κρίση, που είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που εξακολουθούν να είναι πολλά σε ορισμένες χώρες και αποτελούν και κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για τη δυνατότητα των τραπεζών να προσφέρουν πιστώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες. Η αντιμετώπιση της κληρονομιάς που μας άφησε η κρίση είναι ένα θέμα, το άλλο είναι πώς θα φροντίσουμε να μην έχουμε εκ νέου συσσόρευση τέτοιων μη εξυπηρετούμενων δάνειων στο μέλλον. Επ' αυτού λοιπόν σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση επί οδηγίας όσον αφορά τις επιστοτικές ε, οι υπηρεσίε, του αγοραστέ πιστώσεων, του διαχειριστέ πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων. Επίση, προσβλέπουμε στην έναρξη διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον κανονισμό για την ε, ανάκτηση και εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλόμενων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να έχουμε κάποια συμφωνία. Μια άλλη προτεραιότητά μας είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών. Η Κροατία αναγνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πραγματική κεφαλαία ένωση κεφαλαία αγορών και αυτό μπορεί να συνεισφέρει σε πιο σταθερή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με τη, συγχρόνως με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση της ε, Τραπεζικής Ένωσης, πρέπει να έχουμε και μια ρευστή αγορά κεφαλαίων και μια Ένωση Κεφαλαιογορών προκειμένου να ενισχυθεί το ευρώ ακόμα περισσότερο στη διεθνή σκηνή. Και κατά την Προεδρία μας σκοπεύουμε να προσπαθήσουμε να έχουμε νέα μέτρα για να ξεκινήσει μια αναθεωρημένη ε, δράση όσον αφορά την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιογορών. Λαμβάνουμε υπόψη μας το ρόλο που μπορεί να παίξει ο χρηματοπιστωτικός τομέας προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη οικονομία και γι' αυτό σκοπεύουμε να καθορίσουμε προτεραιότητες από ε, αυτού όσον αφορά δηλαδή την Ένωση Αγορών. Επιστρέψτε μου τώρα να στραφώ στο θέμα της φορολόγησης. Το Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα δραστήριο στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια και εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Πολλά θα εξαρτηθούν το κατά πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει έτοιμες νέες νομοθετικές προτάσεις. Οι όροι πράσινοι και ψηφιακή είναι οι λέξεις που είναι πολύ της μόδας, κάθε μέρα τις ακούμε και σίγουρα η φορολόγηση δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση από αυτού του δύο όρου. Εννοείται ότι συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και σκοπεύουμε να διευκολύνουμε τις συζητήσεις και προσβλέπουμε σε προσεχείς δράσεις από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της φορολογίας υπό το φω τη πράσινη συμφωνία. Ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί είναι η ψηφιακή φορολόγηση. Όπω ξέρετε, ο ΣΑ λειτουργεί πάνω σε μια συνολική μεταρρύθμιση για ένα διεθνές ε, σύστημα εταιρικού φόρου προκειμένου να ε, γίνονται λογαριασμοί ψηφιακά. Οι G20 έχουν θέσει ως ε, προθεσμία για μια συνολική λύση το τέλος του 2020 τον, ε, το Συμβούλιο τον Μάρτιο που μας πέρασε αποφάσισε να έχει διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πακέτο φορολογικής, ε, συγγνώμη, ψηφιακής φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέχρι να ολοκληρώσει και ο ΣΑ τις συζητήσεις του. Κατά την Προεδρία μας σκοπεύουμε να στηρίξουμε τις χώρες μέλη στις συζητήσεις αυτές προκειμένου να συμμετάσχουμε και εμείς στις συζητήσεις του ΟΣΑ. Αυτό θα συμπεριλάβει ε, και το θέμα της ε, συμβατότητας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα δούμε τι αντίκτυπος θα υπάρχει στην οικονομία των χωρών μελών και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό τόπο σε όλες τις χώρες ε, μέλη και να προτείνουμε λύσεις εφόσον το περιβάλλον θα είναι κάπως πιο ξεκάθαρο. Εκ παραλλήλου, σκοπεύουμε να έχουμε νέα πρόταση για την κοινή φορολογική βάση για εταιρείε που έχει να κάνει και με τις συζητήσεις μας όσον αφορά την ε, ψηφιακή ε, φορολόγηση. Ανταλαμβάνουμε όμως ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και διάφορα πολιτικά ζητήματα, όπως είναι το πεδίο εφαρμογή. Όσον αφορά το ΦΠΑ, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα το, ποσοστά, τους συντελεστές του ΦΠΑ και την μεταρρύθμισή τους. Πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου όμως να πω και δύο λόγια ή να σας παρουσιάσω ένα από τα θέματα που θεωρούμε εμείς ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις που παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που επηρεάζουν κάποιες από τις νέες χώρες μέλη ιδιαίτερα. Πιστεύουμε ότι οι τάσεις αυτές ελοχεύουν κινδύνους ε, για παράδειγμα όσον αφορά τα δημοσιονομικά των χωρών αυτών και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Η Κροατία λοιπόν έχει αποφασίσει να εισαγάγει μέτρα μετριασμού αυτής της κατάστασης και νέες δραστηριότητες. Εδώ ολοκληρώνω τις αγωγικές μου παρατηρήσεις. Εκ μέρου της ε, Κροατικής Προεδρίας ε, προσβλέπω σε καρποφόρα και αποτελεσματική συνεργασία μας τους επόμενους έξι μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τώρα τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάριτς. Θα δώσω τώρα το λόγο στο, στο, στην πρώτη ομιλήτρια που είναι η κυρία Γιώρη. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και χαιρετίζω και τη δέσμευσή σας και το πρόγραμμα που παρουσιάσετε. Νομίζω ότι η συνεργασία μαζί σας στο επόμενο εξάμεινο θα είναι εξαιρετική γιατί ξέρω πως η καιρή δεν είναι εύκολη, κυρίως για τα όσα έχετε εσείς ε, ξεκινήσει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω και μία ερώτηση στην μητρική μου γλώσσα ε, και να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, στο πρόγραμμα της Κορατικής Προεδρίας έχετε συμπεριλάβει και τα θέματα που άπτονται της δημογραφίας και δίνεται μεγάλη σημασία ε, στις τάσεις αυτές. Η Προεδρία σας λοιπόν έχει σκοπό να προτείνει κάποια μέτρα για να μειωθούν τα αρνητικός δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτής της δημογραφικής τάσης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αυτά τα μέτρα μετριασμού στα οποία αναφερθήκατε. Δεύτερον, θα μπείτε στην ε, ζώνη ευρώ. Ξέρω πώς το σχεδιάζετε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευρώ. Ε, ένα από τα προαπαιτούμενα είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να συμμορφωθείτε με τα κριτήρια αυτά. Και γενικότερα πόσο προετοιμασμένοι είσαστε. Uh, Θα ήθελα λοιπόν και για τις δύο αυτές ερωτήσεις να σας πω πως καταρχήν είναι απόλυτα σχετικές. Η μία δεν σχετίζεται μόνο με την Κροατία, αλλά όπως είπα και προηγουμένως έχει να κάνει με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε οι αρνητικές ε, δημογραφικές τάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τα τελευταία και πιο πρόσφατα χρόνια αλλά νομίζω ότι ε, είναι τάσεις δεκαετίας θα μπορούσα να τις πούμε έτσι με τις επιπλέον πιέσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μέσω μεταναστευτικού και την ολόκληρη μεταναστευτική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν όπως χρειάζεται και αυτό είναι το σκεπτικό ε, πίσω από τις προτάσεις που καταθέτουμε είναι το γεγονός πως εμείς αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερη πρόκληση όπως και τα υπόλοιπα λεγόμενα νέα κράτη. Δεν είναι μόνο η ελεύθερη κυκλοφορία εργατικού ε, δυναμικού, γιατί αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα ε, όταν κάναμε τις εσωτερικές μας ε, εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές αξίες, για την ε, ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία και για τους εργαζόμενους ήταν πολύ σημαντικό το ότι θα μπορούν να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερα. Όμως, όταν βλέπει κανείς πως υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, υπάρχει το brain drain και επιπλέον στοιχεία που συνεισφέρουν περισσότερο στις αποκλήσεις και λιγότερο στις συγκλήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών οικονομιών που είναι και θα έπρεπε να είναι ο βασικός μας στόχος, τότε καιρός είναι να εκφράσουμε το θέμα αυτό και με λόγια. Παράλληλα υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα και κάποιες άλλες συνέπειες αυτών των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, κυρίως στις δημοσιονομικές μας θέσεις και εδώ δεν μιλώ συγκεκριμένα για το ε, πι δέλτα πι και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά και για τους εθνικούς προπολογισμού. Και νομίζω ότι είναι κοινό τόπο ότι το σύστημα περίθαλψης κοινωνικής ασφάλισης ε, συντάξεων αυτή τη στιγμή πιέζονται σημαντικά από αυτές τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις. Είναι πολύ σημαντικό και θα το θέσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών. Σχεδιάζουμε να γίνει ένα άτυπο εκοφήν στο Ζάγκρεμπ 24 και 25 Απριλίου και τα θέματα τα δημογραφικά θα είναι ένα από αυτά τα οποία θα βάλουμε στην ημερήσια διάταξη για να ενθαρρύνουμε τη συζήτηση σε ε, επίπεδο Ευρωπαίων Υπουργών. Τώρα για το ευρώ. Ε, θα κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχω την Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά επειδή μου ζητήσατε ε, απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα της Κροατίας, θα το απαντήσω ε, λαμβάνοντας ε, θέση ως Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας και όχι ως Πρόεδρος της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ξέρετε, πως για μας είναι σημαντικό. Η οικονομία μας εκφράζεται σε ευρώ και έχουμε εκφράσει από πέρσι την ισχυρή μας ε, ε, ε, βούληση να αποτελέσουμε τμήμα του ERM2 σε δύο επιστολές τις οποίες έχει συνυπογράψει ο διοικητής της Εθνικής μας Τράπεζας και εγώ ίδιος και σε επιστολές αυτές δεν α, είπαμε πως είμαστε μόνο πρόθυμοι ε, να μπούμε στον μηχανισμό αλλά ε, να αναλάβουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε λοιπόν απόλυτα δεσμευμένοι στο να παραδώσουμε τα απαιτούμενα ε, σύμφωνα με τα κριτήρια και μόλις μπούμε στον ε, ευρωπαϊκό ε, μηχανισμό ισοτιμιών θα κοινοποιήσουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς πως θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο έτσι ώστε να κινηθούμε προς αυτή την σημαντική για μας διαδικασία γιατί θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία ένταξης ε, στο ευρώ και στη ζώνη Σέγγεν έτσι ώστε να προχωρήσουμε ε, με την ε, ολοκληρωμένη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενημερώσουμε για το σχετικό θέμα αυτό την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ έρχομαι εδώ όποτε μου το ζητάτε και μπορώ να σε εξηγήσω αυτά τα δύο ζητήματα τα οποία για την Κροατία επαναλαμβάνουν ύψη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Λούμα του Σοσιαλιστέ. σοσιαλιστές. Ο κύριος Λούμα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ για την πρώτη Προεδρία της Κροατίας. Είναι πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα σας να είναι χώρα Προεδρίας όπως ε, μόλις ε, βίωσε και η Φιλανδία. Αυτή τη φορά δεν θα αναφερθώ στην ανάγκη μεταρρύθμισης. Οι συναδελφοί μου θα το κάνουν αργότερα. Αλλά θέλω να θίξω ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν αναφέρατε, αλλά που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο και για την Ευρώπη και για τα κράτη-μέλη. Ε, η κατάσταση για την καταπολέμηση ε, της νομιμοποίησης ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η σχετική οδηγία. Ο κ. Ντομπρόφσκης χθε εξέφρασε τις ανησυχίες του για την μη ε, για την ελληπή εφαρμογή της τελευταίας οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Πρόκειται να κινήσει ε, ανέφερε διαδικασίες επί παραβάση κατά κρατών μελών που δεν έχουν ε, θέσει σε ισχύ αυτή την οδηγία και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία του. Υπάρχει ένα πρόβλημα, είπε ο Επίτροπος, ότι ίσως έχουμε το καλύτερο πλαίσιο για την νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο, η Υποφιλανδική Προεδρία, αποφάσισε ότι υπάρχει ανάγκη να σημειωθεί ταχεία πρόοδος στο πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι σημαντικό και όπως καταλάβαμε η Κομισιόν θα προτείνει ένα έγγραφο διαβούλευσης ε, το Μάρτιο φέτος. Εσείς λοιπόν ως χώρα της Προεδρίας στο Συμβούλιο πιστεύω θα μπορούσατε να κάνετε πολλά για να ε, προωθήσετε την ε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας και για να δημιουργήσετε τις συνθήκες μεταρρύθμισης του συστήματος. Αυτό είναι καλύτερο για τους πελάτες, καλύτερο για τις κοινωνίες μας. Οπότε θα να σας ρωτήσω, έχετε τέτοια πρόθεση να ασχοληθείτε με αυτό το σημαντικό ζήτημα του εξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Αξιότιμο μέλος της Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα πράγματι επίκαιρο. Τα είπατε με μεγάλη ακρίβεια. Πρόσφατα, ίσως όχι τόσο πρόσφατα γεγονότα, αλλά σχετικά πρόσφατα, είναι διάφορα γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε καλά και τα οποία αφορούν το ζήτημα αυτό. Αυτό δημιουργεί ανάγκη να δράσουμε όλοι. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως είπατε χθε, ε, είναι κάτι που απασχολεί και τον ε, κύριο Ντομπρόφσκι. Το έχει πάρει πάλι πολύ σοβαρά και αυτός και η Προεδρία και η Επιτροπή. Εμείς ως Προεδρία ήδη έχουμε προγραμματίσει ε, σε επίπεδο ΕΚΟΦΗ να συζητηθεί το Μάιο και τον Ιούνιο το θέμα αυτό στην ΕΚΟΦΗΝ στο ενδιάμεσο έχετε δίκιο. Θα πρέπει να ε, δούμε την έκθεση της Επιτροπής ε, για το στάδιο υλοποίησης ε, της τέταρτης και ιδιαίτερα της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων παρανομής δραστηριότητας. Εγώ ως Υπουργός Οικονομικών θέλω να συνδέσω αυτό το θέμα με το προηγούμενο, επειδή και εσείς αναφέρατε την ε, γενικότερη εμπειρία και προσέγγιση της Φιλανδικής Προεδρίας που εκτιμάμε ιδιαίτερα. Στη δική μας περίπτωση ως κρατική Προεδρία ένα, ε, το θέμα αυτό της καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε, είναι ένα κομμάτι των γενικότερων μέτρων που έχουμε. Δηλαδή εμείς ως χώρα θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό σε εθνικό επίπεδο, αλλά με την εμπειρία που έχουμε εμείς φυσικά και τις γνώσεις που έχουμε και την γενικότερη κατανόηση του ζητήματος αυτού, θα πιέσουμε να γίνουν συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου και αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ανάλογα φυσικά και με τις διαδικασίες όπως τρέχουν στα κράτη-μέλη θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Λέμε βέβαιος ότι τα κράτη-μέλη έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα. Το βλέπω και εγώ από τη δική μου γωνία και από τη δική μου θέση ε, ως Κροάτης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μερικάνο από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρίτσο. Αναλαμβάνετε την προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ σε μια δύσκολη στιγμή με την αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Εύχομαι κάτι ό,τι καλύτερο και η πρώτη σας αυτή προεδρία να είναι επιτυχής. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση. Το ότι θέλετε να επανεκκινηθεί το θέμα αυτό που έχει κολλήσει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι καλό. Ε, συμφωνώ με την εγγύηση καταθέσεων του ΕΝΤΙΣ, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα για τα οποία θέλω να σας ρωτήσω. Πρώτον, το θέμα της έκθεσης σε δημόσιο χρέος, που ξέρετε ότι ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο μέχρι τώρα. Και το άλλο είναι η εξυγένση των τραπεζών. Αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε μία ε, τράπεζα, είναι ότι ο δεύτερος πυλώνας, ο μηχανισμός που έχουμε δηλαδή για την εξυγίανση, δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα και υποθέτω ότι αν είναι αρκετά μεγάλε οι τράπεζε δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και αν δεν είναι απ' την άλλη σημαντικέ, ε, τότε δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Οπότε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, το νομοθετικό πακέτο που εσείς προβλέπετε θα μπορούσε να συμβιβάσει τις ε, διάφορες απόψεις του επιμερισμού κινδύνου ή όχι, τις εγγύησεις καταθέσεων θα δουλέψετε πάνω σε όλα αυτά ή μόνο το θέμα της ασφάλισης θα κοιτάξετε να προωθήσετε. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Ευρωβουλευτά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο ε, μέχρι τώρα συζητιέται εκτενώς στο Eurogroup. Θα λέγω ότι η θέση της Προεδρίας είναι να στηρίξουμε την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και θέλουμε να λειτουργήσει καλά η Τραπεζική Ένωση. Συνεχίζεται το έργο λοιπόν σε επίπεδο Eurogroup, αλλά και σε επίπεδο διαφόρων ομάδων εργασία υψηλού επίπεδου για το ENDIS, την εγγύηση καταθέσεων, και υπάρχει μια συνολική προσέγγιση προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένου στόχου για ένα αποτελεσματικό σύστημα ENDIS. Κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στο να μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση. Αυτό είναι κάτι, ε, πώς να το πω, δεν είναι κανένα μυστικό το έργο για αυτόν τον τρίτο, να τον ονομάσουμε έτσι, πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, βρίσκεται σε κρεμότητα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, υπάρχουν δυσκολίες που βάζετε κι εσείς για το θέμα επιμερισμός κινδύνου ή μείωση κινδύνου, όπως το θέτετε κι εσείς. Η συζήτηση πάντως δεν αγνοεί να ξέρετε τους πρώτους δύο πυλώνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Γιατί παράλληλα με τη δουλειά που γίνεται για το έντις, πρέπει να επικεντρωθούμε και στην εμπειρία που συλλέγουμε και τα μαθήματα που παίρνουμε και τη γνώση που αποκτάμε από τη λειτουργία του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Μόνο έτσι θα ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το πακέτο επιτυχώς στο τέλος. Όσον αφορά λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, την ρυθμιστική δηλαδή αντιμετώπιση της έκθεσης σε δημόσιο χρέος, όλα αυτά αποτελούν μέρος των συζητήσεων που συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδων εργασίας και εμείς ως Προεδρία επίσης θα στηρίξουμε το διάλογο αυτό. Είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη να δώσουμε κίνητρα για τη συνέχιση των ε, συζητήσεων και κάτι που ισχύει και για τις προηγούμενες ερωτήσεις, η θέση της Κροατίας, να ξέρετε ότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε τέτοιες συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων. Κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συζήτηση, γιατί τίθεται στο σωστό επίπεδο η συζήτηση. Κάποιες χώρες μέλη έχουν πει ότι θέλουν να συμμετέχουν στο ΕΡΕΜ, άλλες δεν είναι έτοιμες ακόμα αλλά είναι προς το συμφέρον όλων μας η Τραπεζική Ένωση να λειτουργήσει καλά. Αποτελεί προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιακυλούνες, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας και στη δουλειά που κάνετε, μια και έχετε την προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ. Χαίρομαι για τα σχόλια που κάνατε, για τα δημογραφικά θέματα και για το πώς μπορούν αυτά να ε, μετριαστούν, αλλά θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε μία ε, ερώτηση για την αρχιτεκτονική του συστήματος εποπτείας. Είναι κάπως εκτός πεδίου εφαρμογής της Προεδρίας σας, αλλά μια και είσαστε ε, εδώ και χρόνια στον χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Κροατία, ίσως Έχετε κάποια άποψη για το θέμα της ε, εποπτείας και του συστήματος στην αρχιτεκτονική ε, για την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Πριν από μερικά ε, χρόνια ο κύριος Ντρομπο... μίλησε για τα Twin Peaks που έχουμε από τη μία την προληπτική, το κομμάτι δηλαδή το prudential που είναι σε άλλο σκέλος ε, και αφετέρου την ε, παρακολούθηση και εξού και το Twin Peaks, δηλαδή την δυτή αυτή προσέγγιση. Ξέρω πως η Κροατία είχε κάποια προβλήματα με δάνεια ε, ελβετικών ε, τραπεζών. Είχατε ε, δανειολήπτες, κάποιες δεκάδες χιλιάδες, οι οποίοι προσέφηγαν στις τράπεζες για το θέμα των στεγαστικών δανείων που είχαν πάρει σε ελβετικά φράγκα. Στην FinTech είδαμε ότι υπάρχουν κάποια χρηματοπιστωτικά εργαλεία τα οποία συνεργάζονται με μεγάλες τράπεζες και τα νέα αυτά εργαλεία ενδεχομένω θα δημιουργήσουν μεγαλύτερους κινδύνους ε, για όσου τα χρησιμοποιούν σε μικρέ χώρε κυρίω όπως η δική σας η Λουθινία. Λουθινία. Έχετε λοιπόν αυτό το εποπτικό σύστημα ε, που ε, ονομάζεται Twin Peaks και θα ήθελα να μου πείτε αν το βρίσκεται χρήσιμο ε, και πώς το χρησιμοποιείτε. Επίσης για το επίπεδο δημόσιου δανεισμού στην Κροατία, εφόσον θέλετε να γίνετε μέλος του ευρώ, πείτε μου σε ποιο επίπεδο είναι ο δικός σας κρατικός δανεισμός και πώς έχετε σκοπό ε, να τον αντιμετωπίσετε για την ένταξη στο ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το θέμα της αρχιτεκτονικής, της ε, εποπτείας στο χρηματοπιστωτικό τομέα και όπως είπε και ο αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόσκη, να σας πω πως εμείς ως Προεδρία προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί για οποιασδήποτε δυνητικέ προτάσεις και διάλογο σε συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφερθήκατε εσείς στην περίπτωση αυτή της Κροατίας και των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ελβετικά φράγκα. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και σε, άλλες, ε, και σε άλλα κράτη-μέλη είχαν τέτοιο θέμα. Και από την τελευταία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε πως αυτά τα στοιχεία θα πρέπει ή πρέπει να μας εμπιστοποιήσουν στο πόσο ε, σημαντικό είναι και το κανονιστικό αλλά και το υποπτικό πλαίσιο. Αναφερθήκατε και παραπέμπω στο ότι η πρόληψη ή το ε, προληπτικό σκέλος και τα μέτρα εκεί θα πρέπει να αποτελούν ε, το βασικό μας ε, πεδίο ε, στη σύνταξη όλων των κανονισμών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι υπερβολική η κανονιστική μας δράση. Χρειάζονται και κάποια επιπλέον προηγούμενα μέτρα και γι' αυτό αυτό που θέλουμε να απαιτήσουμε τον τραπεζικό κλάδο είναι να μας επιτρέψει να τα κάνουμε τώρα για τη FinTech είναι ένα θέμα το οποίο θα θέσουμε και στο άτυπο του Ζάγκρεπ. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία μαζί όχι μόνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών να συζητήσουν το θέμα αυτό. Είναι ένα βήμα στο οποίο θα πρέπει να θέτουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι μια νέα πρόκληση η κατάσταση είναι ρευστή και θα έλεγα πως είναι πολύ ταχύες οι αλλαγές. Ε, δεν θα έλεγα επικίνδυνε, αλλά θα πρέπει και η δική μας ε, αντίδραση να είναι ταχύτατη. Για το συγκεκριμένο θέμα του δημόσιου χρέους και πάλι εδώ με, κάποιες, ε, με κάποια εισαγωγικά, γιατί είμαι και υπουργό Οικονομικών της Κροατίας, αν λάβουμε υπόψη τα πέντε κριτήρια τα περίφημα του Μάστριχτ, που είναι τα επιτόκια, ε, η σταθερότητα ισοτιμιών, η, ισότητα, η ισορροπία τιμών και τα δύο ε, δημοσιονομικά κριτήρια που είναι το δημόσιο έλλειμμα, το κρατικό έλλειμμα. Να σας πω πως η Κροατία έχουμε καταφέρει να μειώσουμε και να σταθεροποιήσουμε ε, τα δημόσια οικονομικά μας τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα αλλά συνολικό πλεόνασμα Περιμένουμε βέβαια και τα τελικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν από τον ναι, Eurostat ε, στην, τον Απρίλιο, αλλά για το δημόσιο χρέος τέλη του 2015, να σας πω, πολύ σωστά το είπατε, ήμασταν στο 85% περίπου του ΑΕΠ. Αυτό ήταν ο λόγος και επειδή είχαμε και την, ε, τα μέτρα ανάπτυξης, ε, τα μέτρα της, τα αναπτυξά, αναπτυξά, αναπτυξά, με συγχωρείτε, αναπτυξιακά και επίσης τον εξυγίαση των οικονομικών, ε, να σας πω πως ε, βελτιωθήκαμε πολύ και νομίζω για πέρσι είμαστε στο 71,3%. Περιμένουμε και πάλι τη δημοσίευση των στοιχείων από τη Eurostat. Λοιπόν, αυτά τα 13, 13 ε, ποσοστιαίες μονάδες, όταν τα βάλετε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και των κριτηρίων του Maastricht, θα δείτε πως είναι παραπάνω από ικανοποιητικά και πληρούν τα κριτήρια. Η διάταξη σε αν είσαι πάνω από το 60% η πορεία της μείωσης του δημόσιου χρέους θα πρέπει να είναι τέτοια που θα επιτρέπει να έχει καλύψει το 1 εικοστό τουλάχιστον μεταξύ του τρέχοντος επίπεδου και του 60%. Άρα λοιπόν εμείς μειώνουμε ε, το δημόσιο χρέος στο ΑΕΠ ε, γύρω στο 3% ε, κάθε χρόνο και αν αυτό το δεις ε, με τα όσα έχουμε στις διατάξεις είναι τέσσερις φορές πιο γρήγορα από αυτό το 1,20 ε, το οποίο περιγράφεται. Άρα λοιπόν το δικό μας συμπέρασμα είναι πως ναι, αλλά βέβαια δεν είναι τι θα πούμε εμείς, το θέμα είναι τι λένε οι αριθμοί. Πιστεύουμε πως εκπληρώνουμε το κριτήριο αυτό και στρέφοντας την προηγούμενη ε, ερώτηση, στην αίτησή μας για ένταξη στο ευρώ, εγώ λέω πως δεν μπορούμε να στείλουμε αυτή την επιστολή και να, και να συζητήσουμε το θέμα αυτό εάν δεν εξασφαλίσουμε ε, ε το θέμα, τις επιδόσεις μας στο δημόσιο χρέος κυρίως. Αλλά το τελικό μου μήνυμα είναι μην ανησυχείτε. Εμείς θα ακολουθήσουμε τα σχέδιά μας που είναι και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Το 60% είναι ένα είδος κατόφλι ουσιαστικό αλλά και ψυχολογικό και ελπίζουμε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, που είναι ένας μεσοπρόθεσμος ε, στόχος, να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, από το Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Κροατική Προεδρία. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη απευθύνεται ιδιαίτερα στον Υπουργό. Ξεκινάτε μία διαδικασία ε, προσχώρησης ε, στο ενιονόμισμα η σχέση κόστους-οφέλους αυτής της προσχώρησης ίσως να μην είναι αυτή που ήταν το 2000. Παρατηρώ ότι ορισμένε χώρε εκτό Ευρωζώνη αλλά εντό Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον έχουν καλύτερε επιδόσει από τι χώρε τη Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια. Ποια πλεονεκτήματα λοιπόν αναμένετε εσεί από την προσχώρησή σα στο ευρώ, Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά περισσότερο την κρατική προεδρία. Ε, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον εντελώς αφύσικο αρνητικών επιτοκίων που σε πολλές ε, κυβερνήσεις και πολλούς ενδιαφερομένους ε, γεννά την ιδέα ότι έχει έρθει η ώρα για μαζικές επενδύσεις σε υποδομές να βγούμε από το αυθαίρετο πλαίσιο του 3% του χρέους, ε, του ελλείμματος και ίσως να αναθεωρήσουμε το στόχο του πληθωρισμού του 2% που επίσης είναι αυθαίρετο σε περίοδο αρνητικών επιτοκίων. Ποια είναι η δική σας θέση, η δική σας αίσθηση όσον αφορά την εξέλιξη αυτών των κριτηρίων που είναι τόσο σημαντικά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Και η τελευταία μου ερώτηση προς την Κροατική Προεδρία. Έχουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο με μια αμερικανική πολιτική οικονομικού αθνικισμού ιδιαίτερα επιθετική. Μια μονομερή προσέγγιση σε εμπορικά θέματα χωρίς σεβασμό ούτε νόμων ούτε διεθνών συνθηκών Ποια είναι η θέση τη κρατική προεδρία για το θέμα αυτό, που ούτω ή άλλω θα επιβληθεί στα πράγματα που θα έχουμε να συζητήσουμε στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, πράγματι, το θέμα των ωφελών της προσχώρηση στο ευρώ είναι πολύ σημαντικό. Και εμεί και η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας και η κροατική κυβέρνηση ε, έχουμε προβλέψει το ζήτημα αυτό εδώ και κάποιο καιρό, διότι σε τελική ανάλυση το θέμα δεν είναι απλά να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε μέλη τη ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, να μπούμε στην Ευρώπη και να εισάγουμε το ευρώ απλά γιατί θα εξυπηρετήσει την οικονομία. Θέλουμε μια ενδελεχή ποσοτική ανάλυση όλων των ε, πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων. Μια αναλυση κόστου κόστους-οφέλους, δηλαδή να μην το βλέπουμε μόνο επιφανειακά το πράγμα, αλλά και δυναμικά ποια διδάγματα έχουν αποκομιστεί μέσα από την κρίση, ποια είναι η εμπειρία των σχετικά νέων κρατών μελών που μπήκαν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, το έγγραφο αυτό έχει κυκλοφορήσει το σχετικό έγγραφο ήδη στη χώρα μας, έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, μπορείτε να το βρείτε. Ε, το σκεπτικό ήταν να συνδυάσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση των υπέρ και των κατά. Από δική μας πλευρά, από την πλευρά των κατά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, ειδικότερα στα μάτια των πολιτών μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κροατία ανήκε σε μια ε, πρώην χώρα ενός εντελώς διαφορετικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος και οι πολίτες μας έχουν ζωντανή ακόμα τη μνήμη και τη γνώση της περίοδου υπερπληθωρισμού, υποτιμήσεων κτλ. Οπότε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και δεν παραβλέπουμε τους φόβους τους για το τι θα κοστίσει οποιαδήποτε ε, κρίση, τι κόστος, ε, ποια θα είναι, ποιο θα είναι το τίμημα. Ε, ταυτόχρονα δεν το συγκρίναμε αυτό με την εμπειρία αυτού του κράτους μέλους. Οπότε ποιο ήταν το συνολικό αποτέλεσμα στο θέμα του τιμήματος κατά μέσο όρο μιλάμε για 0,3% ετήσιο πληθωρισμό το πρώτο έτος διότι σε αυτό το συγκεκριμένο για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο μιλάμε ουσιαστικά για μια, ένα αποτέλεσμα πολύ βραχυπρόθεσμο. Δεν θα παραταθεί. Μόλις μπει κανείς στο ευρώ και αλλάξει τις τιμές, ε, ε αυτό συμβαίνει μόνο για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα το κόστος της ε, μετάβασης στο ευρώ, της μετατροπής στο ευρώ, ποιος θα υποστεί το κόστος για τους πολίτες μας είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Ε, σε προηγούμενε ερωτήσει ακούσαμε το θέμα του ελβετικού φράγκου, ε, κατά κύριο λόγο στην Κροατία, πολίτες και εταιρείε έχουν δάνεια είτε σε κούνα ή με κούνα συνδεδεμένη με ευρώ ή σε ευρώ. Παρότι ε, η κούνα είναι το νομισμά μας εδώ και 25 χρόνια, 26. Είναι το εθνικό μας νόμισμα. Όσον αφορά αυτά τα κόστη που είπα ότι θα είναι εφάπαξ, τα ωφέλη ε, είναι πολύ μεγαλύτερα σύμφωνα με την ανάλυση που έχουμε κάνει εμείς. Διότι εν τέλει πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο ε, της συναλλαγματικής ισοτιμίας ε, που θα έχουμε με την εισαγωγή του ευρώ και να λάβουμε υπόψη και τη δομή της οικονομίας μας. Τα νοικοκυριά, τις εταιρείε, το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, σχεδόν όλοι, στους οποίους αναφερόμαστε σχεδόν τα τρία τέταρτα των ισολογισμών τους, έμεσα ή άμεσα έχουν κάπως συνδεθεί στο ευρώ ιστορικά και είχαμε πριν το ευρώ συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με το γερμανικό μάρκο, αλλά υπάρχει μείωση και του πιστοτικού κινδύνου, των κινδύνων για τα επιτόκια. Η Κροατία έχει κάνει πολλά και αυτό μπορείτε να το ελέγξετε και να το διπλοελέγξετε. Αν δείτε τις αποδόσεις των ε, κρατικών μασομολόγων ομολόγων και τα spread ε, των τελευταίων ετών. Ε, τεράστια συρρήκνωση των spread. Παρ' όλα αυτά Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο προόδου σε αυτό το πεδίο, ειδικότερα αν συγκρίνουμε τα δικά μα spread με κάποιε συγκρίσιμε χώρε στη γειτονία μα, στι κέντρο, τις ε, χώρες της κεντρικής και ανατολική Ευρώπη που ανήκουν στο ευρώ. Αυτό λέμε λοιπόν ότι αυτή η ανάλυση ε, κόστου ωφελών δείχνει περισσότερα ωφέλη για την κρυωτική οικονομία. Όσον αφορά την Προεδρία και αυτό που είπατε εσεί για τα αρνητικά επιτόκια, και ορισμένες ε, σκέψεις, συζητήσεις, πρωτοβουλίες ε, για να αλλάξουμε αυτούς τους ε, κανόνες που υπάρχουν εδώ και χρόνια και την οτροπία που έχουμε όσον αφορά το επίπεδο ελλημάτων, πληθωρισμού, τιμών, επίπεδο επενδύσεων κτλ. Θα έλεγα εγώ ότι ένα αναπτυξιακό μοντέλο ενιαίο είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει χωρίς υγιεί σωστές επενδύσεις. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν βιώσιμο. Χρειάζεται λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη τις επενδύσεις, είτε μιλάμε για επενδύσεις, είτε για έρευνα και ανάπτυξη, είτε για οποιοδήποτε είδου επενδύσεις. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός μοντέλου αναπτυξιακού. Παρ' αυτά δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παραβλέψουμε ε, τις, ε, τα αποτελέσματα και τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων των οικονομικών και της δημοσιονομικής θέσης, διότι αυτά είναι στενά συνδεδεμένα. Το ένα εξαρτάται, ή μάλλον θα έλεγα επηρεάζει το ένα το άλλο. Όπως επεσήμανα στην αρχή, ε, η μαλλον θα επηρεαζει το ενα το αλλο οπως επισημανα στην αρχη η κομισιον αυτη τη στιγμή επανεξετάζει πιθανό επανασχεδιασμό των συστημάτων του ΠΑΚ και ΣΥΚΣΠΑΚ η πρωτοβουλία αυτή θα γίνει πιο ευρέως γνωστή το Φεβρουάριο και εμείς ως Προεδρία φυσικά θα υποστηρίξουμε τις συζητήσεις για το θέμα αυτό, διότι τις θεωρούμε πολύ σημαντικές. Και τέλος, όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε και όλα αυτά τα παγκόσμια ζητήματα, ως Προεδρία θα δράσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να ε, ενθαρρύνουμε πρώτα απ' όλα τον διάλογο. Θεωρούμε ότι ο διάλογος έχει πρωταρχική σημασία και φυσικά μέσω του διαλόγου και μια επικοδομητική προσέγγιση ε, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει που θα είναι υποφελεί για όλου. Διότι σε καμία περίπτωση ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι σημαντικό το παγκοσμίο εμπόριο. Ευχαριστούμε. Η ΣΥΑΡ τώρα. Ο κύριος Σούτσικα. Η πρόσφατη συστάση του Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική στην Ευρωζώνη σωστά προτείνει ότι η ενδυνάμει ανάπτυξη παραμένει χαμηλή και κάτω από τα επίπεδα πρώτης κρίσης και υπάρχει κίνδυνος η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει μία περίοδο με χαμηλή παραγωγικότητα και μεγένθηση. Πολύ συζητάμε τώρα για την Πράσινη Συμφωνία. Όμως, βραχυπρόθεσμα, αυτό μπορεί να σημαίνει παραπάνω δαπάνες, χωρίς όμως να έχουμε παραπάνω ε, παραγωγή, μια που υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα. επίγει λοιπόν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν γρήγορα και να πιέσουμε ώστε να επανέλθουν τα επίπεδα ανάπτυξης στα επίπεδα πρώτης κρίσης. Συχνά οι συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αγνοούνται και το Συμβούλιο Παραγωγικότητας δεν έχει αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων. Η Ισπανία, για παράδειγμα, θα κάνει πίσω ε, σε σχέση με μεταρρυθμίσεις για τα εργασιακά που είχε οθετήσει η δικιά μου η χώρα, η Σλοβακία πάλι, βλέπει την κυβέρνηση να καταστρέφει διάφορα μέτρα βιωσιμότητας. Οπότε ρωτάω εσείς πώς θα βελτιώσετε την, τα κίνητρα που έχουν οι χώρες μέλη ώστε να επιταχύνουν ε, τις μεταρρυθμίσεις και να μην αντίθετα τις ανατρέπουν. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά προσπαθήστε παρακαλώ να το πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη Ευρωβουλευτά. Θα έλεγα ότι με την ερώτησή σας δεν κάνετε απλώς μια ερώτηση, ε, ουσιαστικά θέλετε και την απάντηση γιατί όταν θέτουμε το θέμα της ενδυνάμει ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, πάντα έχουμε την δυσκολία να βλέπουμε ότι τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από εκείνα που είχαμε πριν την κρίση. Θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και όλοι πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα επίπεδα ζωής, τους μισθούς στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μας αφορά όλους και μπορούμε να το δούμε και κανονιστικά. Αλλά από την άλλη οι μισθοί και οι δαπάνε έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Έτσι είναι η συνάρτηση της ανάπτυξης. Τώρα, η δημοσιονομική πολιτική των χωρών μελών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε να ε, προχωρήσει και σε ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η σωστή ερώτηση βέβαια είναι πώς να δώσουμε κίνητρα. Πώς να είναι πιο ελκυστικές αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γιατί ξέρουμε ότι ε, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αλλαγές και πάντα υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικής οικονομίας εδώ πέρα που παίζει. Οπότε εκτιμούμε πάρα πολύ που θέτεται το θέμα αυτό ε, του προγράμματος επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Το είπα και στις αγωγικέ μου παρατηρήσεις ότι από τη μια έχετε το στοιχείο αυτό των μέσων προπολογισμού για την ε, σύγκληση και από την άλλη μεριά σε θελεντική βάση αναχώρα ε, για τις χώρες μέσα στο ευρώ αλλά και για τις άλλες που δεν συμμετέχουν στο ευρώ. Υπάρχουν ε, μέτρα που δίνουν κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και για επενδύσεις. Οπότε, εφόσον έχουμε μια κοινή προσέγγιση, μπορούμε να βοηθήσουμε στη συνειδητοποίηση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ότι χωρίς κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα δεν μπορούμε να περιμένουμε αύξηση στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Μιλάμε για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή την εποχή αλλά θα έλεγα ότι το θέμα της δυνατότητας ανάπτυξης πηγαίνει και πέρα από αυτήν την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ πάντως για την ερώτησή σας και κυρίως για το ότι μέσα από αυτή την ερώτηση δίνεται και την απάντηση. Πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση της πολιτικής ελίτ και όλων των χωρών μελών, ώστε να προχωρήσουμε συνολικά και να καταλάβουν και οι πολίτες ότι είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστούμε, Μούρεσαν. Ελκ τώρα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας συγχαρώ για το βιώσιμο τρόπο με τον οποίο υπό την ηγεσία της κυβέρνησής σας η οικονομία της Κροατίας ε, αναπτύσσεται μειώνοντας το δημόσιο χρέος με τον τρόπο τον οποίο εξηγήσατε, με σταθερή ανάπτυξη και όλο και χαμηλότερα ε, ποσοστά ανεργίας. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, για το ε, μέσο του προϋπολογισμού για την σύγκληση και για την ανταγωνιστικότητα. Γίνανε πάρα πολύ περίπλοκες συζητήσεις εδώ για το πεδίο επαρμογής, για το εργαλείο, για τη διακυβέρνηση και διαχείριση αυτού. Σας ρωτώ λοιπόν, χρηματοδότηση αυτού του μηχανισμού. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε φιλόδοξα εργαλεία, τότε θα πρέπει και η χρηματοδότηση να επαρκεί. Γνωρίζουμε όλοι ποιε είναι οι προτάσεις που έχει κάνει ε, στο ΠΔΠ η Φιλανδική Προεδρία. Εσείς ποιο θεωρείτε πως είναι το κατάλληλο ε, επίπεδο χρηματοδότησης για αυτά τα δύο εργαλεία. Επίσης, πότε αναμένεται να γίνει μια συμφωνία, να βρεθεί μια συμφωνία για τα δύο αυτά εργαλεία στα πλαίσια των, του συζητήσεων για το ε, ΠΔΠ. Και δεύτερον, για το νέο Green Deal. Μιλήσατε για το γεγονός πως πρέπει να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θεωρείτε πως θα λειτουργήσει και επίσης ο δίκαιος μηχανισμός ε, μετάβασης ποιο είναι ο τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, πόσο φιλόδοξοι πρέπει να είμαστε ε, σε όγκο χρηματοδότηση, αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκούν και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη να υποστηριχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα συγκεκριμένα κομμάτια του προγράμματος ε, και των εργαλείων που αναφέρατε, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των συζητήσεων που γίνονται για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές και η Προεδρία για το θέμα αυτό, όπως και για άλλα που σχετίζονται όχι μόνο με τούτο, αλλά ε, ευρύτερα με τις ΠΔΠ, περιμένουμε για την πολιτική... Ε, κατεύθυνση και πλαίσιο που θα ε, δημοσιευθούν ε, σύντομα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε κάποια δέσμευση, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο, αλλά για σας που είστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας, το σημαντικό είναι να ξέρετε πως είμαστε ε, έτοιμοι και θα είναι ένας ολόκληρος καταράχτης ε, δράσεων, τεχνική εξέταση άστρο κατά άστρο κτλ. Θα ξεκινήσουν αμέσως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, μόνο αυτό έχω να απαντήσω. Για το Green Deal χτες κάναμε το πρώτο κοφήν της χρονιάς. Το συζητήσαμε. Ε, πρέπει να σας πω που η συζήτηση ήταν εξαιρετικά επικοδομητική, καρποφόρος, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν ανταλλάξει μεν απόψεις, αλλά θεωρώ πως είναι σωστό αυτή τη στιγμή που ξεκινά η νέα εντολή να έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα μπροστά μας και όπως είπα και χθες, να το συζητήσουμε όχι μόνο μήνες, αλλά και χρόνους, έτσι ώστε να καταλήξουμε μια επιτυχή σφαιρική συμφωνία. Εμείς, ως Προεδρείο, το είπαμε και χτες και θα το επαναλάβω και σήμερα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να συμμετάσχουμε, να οργανώσουμε όσο διάλογο χρειαστεί σε τεχνικό επίπεδο στο Συμβούλιο ή αλλού, έτσι ώστε να δώσουμε μια σωστή απόκριση σε όλα τα ερωτηματικά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τάγκ από τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και καλή τύχη για το εξάμεινο αυτό. Αναφέρατε στην έκθεση κατά χώρα και ξέρουμε ότι η Αυστρία άλλαξε τη θέση της και τώρα θα υπάρχει δική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Η Φιλανδική Προεδρία ήδη έχει κάνει άλλη πρόταση λαμβάνοντα υπόψη τις ε, συστάσεις τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και αυτό θα διευκολύνει τη συζήτηση για τη νομική βάση της πρότασης. Δεδομένων αυτών θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία να ξανασυζητηθεί στην ε, ατζέντα αυτό το στοιχείο, ειδικότερα καθώς τώρα υπάρχει ένα τέμπλετ, ένα πρότυπο για τις εκθέσεις αυτές και νομίζω 20 μεγάλες εταιρείε ήδη το έχουν υιοθετήσει, οπότε πρέπει να βιαστείτε, θα έπρεπε να πω ποια είναι τα βήματα λοιπόν που προτίθεστε να κάνετε για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, έχει συζητηθεί αυτό και στο ECOFIN πρόσφατα. Thank you, honorable. Uh, Ευχαριστώ πολύ αξιότιμο μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, το θέμα ε, συζητήθηκε ξανά πρόσφατα αν δεν ε, έχετε πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ούτω ώστε να κατανοήσουμε όλοι γιατί μιλάμε, οι εθνικές φορολογικέ αρχές ήδη ανταλλάσσουν πληροφορίε για τις ε, εταιρείε σύμφωνα με την οδηγία διοικητική συνεργασίας. Ωστόσο, το ζήτημα τώρα που συζητείτε ξανά είναι η κρατική προσέγγιση αυτών των συγκεκριμένων δεδομένων. Όπως ξέρετε, η εργασίες σε επίπεδο Συμβουλίου έχει έχουν προχωρήσει αλλά λόγω αυτής της νομικής βάσης ε, που είναι επίμαχη προφανώς εμείς ως Προεδρία θα πρέπει να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες για να υπάρξει στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και να μπορέσουμε έτσι να προσδιορίσουμε πιθανές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε με αυτό το αρχείο. Αλλά σήμερα και θα το γνωρίζετε κι εσείς ε, από τη θέση που βρισκόμαστε έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου ε, υπάρχει, είναι επίμαχο ζήτημα αυτή η νομική βάση και το πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά όπως είπα θα εστιαστούμε ιδιαίτερα στο διάλογο με τα κράτη-μέλη και με τα θεσμικά όργανα ώστε να βρούμε μια λύση η οποία όπως είπα να βοηθήσει την ε, κατάσταση να προχωρήσει δευτερολογία του κύριου Τάν. Ξέρετε, στη δική μου χώρα, στις κατοχώρες, ο άσποδος εχθρός μου είναι η ΣΕΛ, η εταιρεία αυτή, η οποία πραγματοποιεί εκθέσεις κατά χώρα στα λογιστικά της βιβλία και ξέρουμε ότι δεν πληρώνουν φόρο ως εταιρεία στις κατοχώρες. Ε, θα επέρχονται αλλαγέ, επίκεντα αλλαγέ πιστεύω. Έρχεται η ώρα. Όταν λέτε θέλετε να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη, τι εννοείτε θα ε, πιέσετε, θα σημειώσετε κάποια επιτυχία μέσα στο επόμενο εξάμεινο ή απλά θα ξανακάνετε τις βασικές ε, εργασίες. Όπως είπα, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα της νομικής βάσης δεν έχουμε εμεί τέτοια δυνατότητα. Ούτε εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε, να δικάσουμε ή να ε, λάβουμε κάποια τελική απόφαση. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η διαφορετική κατανόηση των άρθρων τη συνθήκη, εμεί μπορούμε να πιέσουμε για να γίνει ο διάλογο. Διότι, όπω είπα, αναμφίβολα γνωρίζουμε το γεγονό αποτελεί κομμάτι ε, τη δέσμη μέτρων που έχουμε εμεί αυτή τη στιγμή προβλέψει για το Συμβούλιο εδώ και καιρό το συνολικό ε, επίπεδο της φορολόγησης και ειδικότερα σε επίπεδο BEPS και όσα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι των συζητήσεών μα και των διαλόγων μα πώ θα βελτιώσουμε τη συνολική εταιρική φορολογία παγκοσμίω. Όχι μόνο για τι εταιρείε Ευρω... που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στα κράτη τη, αλλά και πέραν αυτών. Ε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε ω Προεδρία. Ευχαριστούμε. Βίλικα από το Ρινιού, παρακαλώ, ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ κάθε επιτυχία στην κρατική Προεδρία. Έχω μια ερώτηση για το σύμφωνο ε, σταθερότητας. Ε, προβλέπετε μια αναθεώρηση, η Επιτροπή θα μας την ανακοινώσει στα τέλη αυτού του μήνα από ό,τι φαίνεται και στην επόμενη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ προφανώς θα συζητηθούν οι παράμετροι της ε, αναθεώρησης αυτής. Το θέτω αυτό στα πλαίσια τη δικιά σα προεδρία και τη φιλοδοξία σα να έχουμε μια Ευρώπη που αναπτύσσεται αγωνίζονται οι οικονομίες της Ευρώπης. Η μεγέθυνσή μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι με τις επιπτώσεις, τις γνωστές, στην απασχόληση, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση κλπ. Οπότε, όσον αφορά την αναθεώρηση αυτή καθ' αυτή, μιλάμε για τη σταθερότητα, αλλά δεν δίνουμε αρκετή σημασία στην ανάπτυξη. Όταν γίνει λοιπόν αυτή η αναθεώρηση θα είναι αμερόληπτη, θα αναλύει σε βάθος τις επιπτώσεις, τον ε, αντίκτυπο που έχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, στις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά και από πλευράς των οικονομιών πώς θα μπορέσουν να επενδύσουν όχι στο σημερινό περιθώριο που υπάρχει, ε, κύριε Υπουργέ, αλλά ε, σε υποδομές, ε, εκπαίδευση, υπηρεσίες κλπ. κλπ. Πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα στις οικονομίες και από πλευράς του κεφαλαίου. Και όχι και ομάδες, αλλά το λέω προσωπικά, ότι Εμένα με απασχολεί πολύ. Φοβάμαι ότι θα αποτελέσει στενό κορσέ στις εθνικές οικονομίες και δεν θα μπορούν να επενδύσουν με τι κεφαλακέ ε, απαιτήσει που υπάρχουν. Αλλάζει η δημογραφία με τραγικό τρόπο στην Ευρώπη, γερνάμε και θα έπρεπε να μπορούμε να σχεδιάσουμε για τα ενδεχόμενα που μας περιμένουν. Οπότε εσείς θα χρησιμοποιήσετε την Προεδρία σας ώστε να διασφαλίσετε πως κάθε ανάλυση που γίνεται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα λαμβάνει υπόψη ευρύτερες παραμέτρους, όχι μόνο την νομισματική πολιτική και τις κυβερνητικές δαπάνες, αλλά και γενικότερα τον αντίκτυπο στις επενδύσεις ευρύτερα στην ε, Ευρωζώνη και τις οικονομίες της. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, Μαξιότιμη Ευρωβουλευτέ συνδέει τη ερώτησή σας με μία από τις προηγούμενες. Και έτσι θα επαναλάβω και εδώ αυτό που είπα πριν, ότι δηλαδή ακριβώς αυτό είναι ένα από τα ζητήματα κλειδί που πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε. Το είπα και στις αγωγές μου παρατηρήσεις ότι έχουμε κάποια μεγένθηση, η οποία όμως επιβραδύνεται από το 2018 και μετά. Επίσης, μαθαίνουμε ε, τα μαθήματά μας, παίρνουμε τα μαθήματά μας από τις προηγούμενες κρίσεις και νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε υπόψη και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να απαντήσω ε, σε κάποια από τα ερωτήματά σας για το τι θα περιλαμβάνει η έκθεσή τους. Θα το δούμε το Φεβρουάριο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε διάλογο επ' αυτού. Τον Απρίλιο Πάντως υπάρχει άτυπο εκοφήν στο Ζάκρεπ και θα βάλουμε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη για να συνεχιστεί ο διάλογος. Πάντως όλα τα στοιχεία που θέτετε εσεί είναι σωστά. Η οικονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, αλλά δεν φτάνει. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις επενδύσεις, όχι μόνο τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές, στις διάφορες ε, χώρες και στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά υπό το φως της εμπειρίας που έχουμε από τη δημοσιονομική κρίση, δεν πρέπει να γνωρούμε ε, στοιχεία και αποτελέσματα της οικονομικής αυτής κατάστασης. Οπότε το πακέτο των 2 και των 6 οδηγιών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θυμάμαι εδώ και άλλες συζητήσεις παλιότερα που είχαμε στο Συμβούλιο που είχαμε θέσει και το εξή. Πρέπει να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τους άλλους, αλλά να διαπαιδαγωγήσουμε και τους πολίτες μας, ότι δεν πρόκειται μόνο για μια χρονιά ανάπτυξη, τι ποσοστά έχουμε κτλ. Όχι, είναι γενικότερο. Πρέπει να ενισχυθεί και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, η δυνητική. Και Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας σε εσάς, αλλά και τους προηγούμενους, γιατί πράγματι παράλληλα με τη διαδικασία αυτή πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει όθηση στη δυνατότητα μεγένθησης που μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη. Πάντως και εγώ προσβλέπω σε αυτήν την ε, αναθεώρηση και τον ανασχεδιασμό ε, ε, των ε, ρυθμίσεων ε, του πακέτου των δύο και των έξοδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσρα Μαλτεκένε, ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για τις απαντήσεις και θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας πω το εξής. Όταν μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα της Προεδρίας σας, ανακοινώσατε που θέλετε μια ισορροπημένη και βιώσιμη συμφωνία για τις ΠΔΠ. Στην συνθήκη η συνοχή και η ΚΑΠ είναι κοινέ πολιτικές και δυστυχώς έχουμε και νέες προκλήσεις οι οποίες όμως και αυτές χρειάζονται χρηματοδότηση ε, που δεν θεωρούνται κοινέ πολιτικές, κοινωνική, η πολιτική ασφάλειας, η πολιτική παιδείας και μα είπατε πως η μακροπρόθεσμη πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην σφιχτή δημοσιονομική ε, πειθαρχία και στην χρηματοδότηση των στόχων μας. Καλά όλα αυτά. Όμως οι στόχοι που έχει η ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιτυχθούν μόνο αν αυξήσουμε τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να βρεθεί επιπλέον χρηματοδότηση ή αν κάνουμε μία αναδιανομή των ε, κονδυλίων έτσι ώστε από την ΚΑΠ να πάρουμε πόρους για θέματα όπως η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή στην Λιθουανία έχουμε ε, ιδιαίτερα δυσαρεστημένες μερίδες πληθυσμού που μειώνονται τα γεωργικά κονδύλια και τα λόμπι των γεωργών είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη. Ακούγονται, επηρεάζουν, είναι ορατοί. Στα νέα κράτη-μέλη, στην Ανατολική Ευρώπη, είναι και ε, ε, εξαιρετικά κομματικοποιημένοι έχουν πολιτική δράση, άρα λοιπόν ρωτώ, θα καταφέρετε να επιτύχετε τους φιλόδοξους στόχους σας και πιο συγκεκριμένα. Θα στηρίξετε ρεαλιστικές θέσεις και θα πετύχετε συμφωνία ή θα ακολουθήσετε τις αρχές σας και θα στηρίξετε τι μεταρρυθμίσει που ανακοινώνετε, οι οποίε κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο φιλόδοξε όσο θα μπορούσαν να είναι. Thank you very much, uh, of the Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που κάνατε. Η απάντησή μου έχει να κάνει και με τη μεταρρύθμιση ε, και θα επαναλάβω τα όσα είπα και για τα προηγούμενα ζητήματα. Και σε αυτούς τους τομιακούς ε, κλάδους του, των ε, ε, ΠΔΠ είμαστε στη φάση της συζήτησης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και σίγουρα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα μιλήσουν για τα συγκεκριμένα ζητήματα σαν αυτά τα οποία εσείς αναφέρατε. some kind final proposal and the guidance. Και εκεί θα μας κατευθύνουν έτσι ώστε να δούμε ποια τακτική θα ακολουθήσουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς η Προεδρία θεωρούμε πως το σημαντικό για εσάς είναι να γνωρίζετε πως εμείς είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι, απόλυτα έτοιμοι για όλα τα επόμενα βήματα εφόσον λάβουμε τις πολιτικές μας οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα έσοδα. Δεν ξέρω αν θεωρείτε εσείς την μεταρρύθμιση του συστήματος ίδιων πόρων ή είχατε κάτι άλλο κατά νου. Νομίζω όμως ότι η απάντησή μου καλύπτει και τούτο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρικ Βερκά από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Η Υπουργέ ευχαριστω πολυ ο Μάρικο απο τους σοσιαλιστες ευχαριστω ήδη το ζήτημα της Τραπεζικής Ένωσης, η, με μεγαλύτερη ακρίβεια της ενίσχυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στο επίκεντρο του ζητήματος ε, βρίσκεται το σημερινό αδιέξοδο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων. Και η ερώτησή μου είναι, σκοπεύετε να προσπαθήσετε να βρείτε ενέσιδες ιδέες για να βγούμε από αυτό το διέξοδο, για να γίνει μια νέα μεγάλη, να γίνει ένας νέος μεγάλος συμβιβασμός μεταξύ των χωρών που θέλουν να αμοιβαιοποίηση του κινδύνου και εκείνων που θέλουν μείωση των κινδύνων. Έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα πρέπει να προχωρήσετε ή πού θα αναζητήσετε νέες ιδέες για αυτό το ζήτημα. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά πιο συγκεκριμένα την Κροατία. Βλέπω θετικά την απόφαση της Κροατίας να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Ένα από τα κριτήρια είναι να μπει κανείς για δύο χρόνια στο σύστημα ERM2. Η εικόνα είχε ουσιαστικά συνδεθεί με το ευρώ και αυτό δεν θα μπορούσε να... Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι γιατί οι κανονες ε, erm ERM2 προβλέπουν κάτι διαφορετικό ε, για ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν φοβάστε λοιπόν ότι εντός ε, της ERM2 θα έχετε μεγαλύτερη αστάθεια της, του νομισματός σας. Thank you. Thank you, of the... Ευχαριστώ αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε για το ίδιο και την περαιτέρω εμβαθύνση της Τραπεζικής Ένωσης. Κάποια πράγματα που είπα ήδη ήταν ότι θα είμαστε παρόντες σε αυτό το διάλογο σε επίπεδο Eurogroup μαζί φυσικά με το Συμβούλιο ούτως ώστε όπως είπατε πολύ σωστά να βγούμε από αυτό το αδίέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ε, ωστόσο στο ενδιάμεσο ε, και ε, θα επανεξετάσουμε τους δύο της Τραπεζικής Ένωσης και την επιπλέον πρόοδο που όλοι αναμένουμε για το είδης. Η κατάσταση λοιπόν έχει ότι είναι, χρειάζεται αμοιβαία κατανόηση ε, της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, οπότε ο διάλογος θα συνεχιστεί. Όσον αφορά το ευρώ σε σχέση με την κούνα, το εθνικό μας νόμισμα και το ERM2, το μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας 2. Έχετε δίκιο ε, για αυτά που είπατε για την Κροατία και την Εθνική μας Τράπεζα και η γενική συναλλαγματική πολιτική δεν είναι μόνο των τελευταίων δύο ετών, αλλά ξεκίνησε το 1993-1994 με την εισαγωγή της Κούνα. Έχουμε ε, κειμενόμενο επιτόκιο, ε, κειμενόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, όπως είχατε πει, και συνδέεται η εικόνα παλιότερα με το γερμανικό μάρκο και σήμερα με το ευρώ. Οπότε αυτές ε, οι ευξομοιώσεις ε, τι τελευταίε δυόμιση δεκαετίε ήταν περιορισμένες. Ο διάλογος που είχαμε με την Εθνική Τράπεζα και φυσικά η Εθνική Τράπεζα είναι αυτόνομη ε, αρχή εποπτεία στην Κροατία αλλά σε δημόσιες τους δηλώσεις λένε ότι παρότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να τολμήσει κανείς να αναφέρει συγκεκριμένα νούμερα όσον αφορά τη συνεργαματική ισοτιμία τη στιγμή της εισαγωγής. Δεν αναμένεται κάποια τεράστια διαφορά ε, στην αξία της κούνα. Ε, πολλές φορές έχουμε ξαναδεί και πριν από την ε, περίοδο της ύφεσης έχουμε δει να υπάρχει κάποια σημαντική απόκληση μέσα στο πρώτο έτος, ειδικότερα ε, το, την θερινή περίοδο λόγω της εισαγωγής συναλλάγματος. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις ε, στην κούνα σε αντίθεση με το υπόλοιπο του έτους, όπου ε, ηρεμεί λίγο η διαδικασία παρά τις ε, όποιε προσδοκίες, τα πράγματα δεν άλλαξαν ιδιαίτερα στην περίοδο της ύφεσης, ούτε έχουν αλλάξει σήμερα. Οπότε η Κρατική Εθνική Τράπεζα ε, υιοθετεί ενεργά κάποια μέτρα και εργαλεία ανοιχτή αγοράς, ούτω ώστε να ε, προσπίσει τη σταθερότητα αυτή και ειδικότερα με την εμπειρία που έχουμε και τη γνώση που έχουμε δεν αναμένουμε τεράστιες αυξομοιώσεις στο, κατά την είσοδο στο ERM2. Ευχαριστούμε. Α, έχετε συμπληρωματική. Δέκα δευτερόλεπτα. Ήθελα να τονίσω ότι στην περίπτωση της Κροατίας η απέτηση αυτή για είσοδο στο ERM2 δεν έχει νόημα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ε, τώρα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ε, μιλήσουμε για πιο περίπλοκα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς τα οικονομικά είναι περίπλοκα, αλλά πρόκειται και για τη δημογραφία. Οι εξελίξεις είναι ανησυχητικέ. Έχουμε και το θέμα της εξωτερικής μετανάστευσης, τις συγκρούσεις που αναφέρονται πολύ. Αλλά χώρες όπως είναι, Κροατία, Λετωνία και άλλες, ε, διαπιστώνουν ότι έχουν όλο και λιγότερο ενεργό πληθυσμό με επιπτώσεις σημαντικές στη δημοσιονομική τους κατάσταση και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ε, των οικονομιών τους, της αναπτυξής τους κτλ. Η Κροατία είπατε ότι θα προτείνει, ίσως ήδη το έχετε προτείνει, διάφορα μέτρα μετριασμού του φαινομένου και δραστηριότητες. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Έπειτα, σε σχέση με το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Υπάρχουν σχετικά νέες χώρες, ίσως όχι η Κροτία, άλλες, να διαπιστώσουν μειώσεις στα διαρθρωτικά τους κονδύλια, συνοχή κλπ. Σε σχέση λοιπόν με τις δημογραφικές τάσεις που θα συνεχιστούν, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και αν σε μερικές χώρες υπάρχουν κάποιες αλλαγές, μια μικρή αύξηση για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ίσως κάποιες από αυτές τις χώρες να βρεθούν ε, σε αδιέξοδο. Η απώλεια των κονδυλίων με τις αλλαγές της παραμέτρου χρηματοδότησης θα μπορούσαν να δημιουργούσουν πραγματικά οικονομικά προβλήματα. Οπότε με τριασμός, δραστηριότητες μπορείτε να επεκταθείτε περισσότερο. Ευχαριστώ αξιότιμη Ευρωβουλευτά. πολύ σωστά αναγνωρίζετε το πρόβλημα το δημογραφικό μεταξύ άλλων και δεν πρόκειται μόνο για τη δικιά σας χώρα, όλες οι βαλτικές χώρες αλλά και άλλες όπως και η Κροατία προσπαθούμε ατομικά σε εθνικό επίπεδο δηλαδή να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις ιδιαίτερα στο δημογραφικό. Η λογική πάντως για μας που θέτουμε το θέμα σε επίπεδο Συμβουλίου είναι ότι προφανώς και χρειάζεται να υπάρξει μια κοινή κατανόηση του προβλήματος. Δεν λέω ότι με τον ίδιο τρόπο το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά πάντως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει το μαγικό ραβδί ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο Ευρώπης που να λύσει αμέσως το ζήτημα. Εγώ θα έλεγα ότι οι δημογραφικές προκλήσεις και αν τις συνδυάσουμε και με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν να κάνουν, με τις ασφαλίσεις, τα εξοδοτικό κτλ, οδηγούν στο να θέλουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση και τη συνδυτοποίηση ακόμα περισσότερο ότι χρειάζονται ε, διαρθρωτικές αλλαγές και ίσως προσαρμογή των συστημάτων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν για να επανέλθω στο θέμα της ε, δυνητικής ανάπτυξης, χρειάζεται νέα απασχόληση, μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία αποτελούν την απάντηση ε, στο όλο ζήτημα. Η λογική, η δικιά μας, που μας οδηγεί να θέσουμε το θέμα στο Συμβούλιο, είναι ακριβώς λοιπόν όλα αυτά και γενικότερα στο χαρτοφυλάκιο υπάρχει το θέμα το δημογραφικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς από πλευρά του Συμβουλίου θα δώσουμε επίσης όθηση στο ζήτημα για να στηρίξουμε τη χώρα σας αλλά και άλλες χώρες αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί λίγο πολύ όλες τις χώρες. Ευχαριστούμε. Catch the ο Ρόμπερτ Βίλαντ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπω και που είμαι σε αυτή την αίθουσα και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Υπουργό από την Κροατία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο καλά ξέρετε το θέμα σας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συχνά έθετα σε αυτές τις συνεδριάσεις είναι η ζημιογόνος επίπτωση των αρνητικών επιτοκίων στην Ευρώπη, στον κλάδο της αποταμίευσης, που αποτελεί ένα τεράστιο ε, πλεονέκτημα για μας. Επίσης, ανησυχώ ιδιαίτερα για τα αρνητικά επιτόκια και για το πώς επηρεάζουν το καπιταλιστικό σύστημα και του μηνύματος που στέλνουν γιατί ξέρετε ότι είναι το κόστος του χρήματος που ε, ορίζει το πώς θα πάει το καπιταλιστικό σύστημα. Οπότε εδώ έχουμε τα εξής δύο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να προχωρήσουν σε διακανονισμούς οι εταιρείε με αποτέλεσμα να γίνονται εταιρείε ζόμπι όπως ε, στην Ιαπωνία και επιπλέον ε, δεν έχουν κάποιο ε, κίνητρο για να δανείζουν οι τράπεζες γιατί είναι αρνητικά τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περιορισμένη χρονική στιγμή που έχουμε μια τελείως αντίστροφη τάση, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία κινητής ή ακίνητης περιουσίας έχουν εκτιναχθεί είναι ε, μια φούσκα που δημιουργείται. Εγώ δουλεύω στο τραπεζικό σύστημα και θα επιστρέψω σε μια εβδομάδα στην επενδυτική τραπεζική μου δραστηριότητα και ακούω πάρα πολλά έξυπνα σχόλια από ε, μέλη της ομάδας ECR, από την IG για την Τραπεζική Ένωση, για την ασφάλεια των καταθέσεων και την ασφάλιση αυτών. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στον... Ε, ε, ευρωπαϊκό μηχανισμό έχουμε γύρω στα 55 δις. Εάν έχουμε νέο, νέα κρίση, φτάνει. Και τι μπορεί να κάνει κανείς για να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια ενδεχόμενη κρίση. Γιατί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουμε ο κοντι νότερος μας γείτονες να περάσει μια κρίση σαν το 2008 όπου είχαμε οικονομικά σοκ, ε, ε, ύφεση από πληθωρισμό φρικτά για μικρά κράτη όπως η Κροατία. Οπότε για μένα και για τη χώρα μου πιστεύω πως θα έπρεπε η Ευρώπη να μην είναι υπερεξαρτημένη από την νομισματική πολιτική τώρα που είναι αρνητικά τα επιτόκια. Και σας λέω το εξής, στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση τα επιτόκια ήταν στο 4-4,5%. Οπότε υπήρχε περιθώριο να μειωθούν. Όταν όμω έχει αρνητικά επιτόκια, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει να τυπώσει χρήμα. Και να τυπώσει χρήμα είναι μία, ε, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου, ε, τρελή παρόρμηση, ε, χωρί αποτέλεσμα και ελπίζω πω αυτά τα ζητήματα θα κοιτάξετε. Είναι ερωτηματικά που μου προκαλούν ανησυχία και θα ήθελα να μου πείτε, εσεί τώρα που θα έχετε την Προεδρία του Συμβουλίου θα προωθήσετε αυτό το οποίο εγώ ε, ονομάζω μια επιλογή ελεύθερης αγοράς, δηλαδή λύσεις όπως περισσότερος ανταγωνισμός, ε, μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην, ε, στο χώρο της ε, προσφοράς, κίνητρα για επενδύσεις και να επιτρέψετε περισσότερη ανάληψη κινδύνων. Γιατί με το νέο Green Deal και το τελευταίο που έχω να πω, αυτή τη στιγμή εξαρτώμαστε ιδιαίτερα από, τον, ε, από μηχανής Θεό, ο οποίος θα διορθώσει την εξαιρετικά αργή ανάπτυξη στην Ευρώπη και με ανησυχεί. Δηλαδή, φοβάμαι πως βραχυπρόθεσμα, όπως και στην γερμανική αυτοκίνητο βιομηχανία που χάθηκαν 40.000 θέσεις εργασίας, αυτές οι πράσινα, αυτά τα πράσινα project θα ε, μας πλήξουν περισσότερο ε, βραχυπρόθεσμα και μετά ενδεχομένως κάτι θα προσφέρουν. Σας ευχαριστώ, μου δώσατε 3 λεπτά και 45 δεύτερα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Δύο λεπτά όμως για την απάντηση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομο. Εντάξει, το δικό σας ε, υπόβαθρό το και το ε, επαγγελματική στραστιδομία φαίνονται από την ερώτηση. Θα απαντήσω ένα τμήμα της ερώτησης ως Υπουργό Οικονομικών της Κροατίας που ανέλαβε αυτή τη θέση μια εποχή που η Κροατία ήταν πάνω από 300 μονάδες βάσης στα spread για τα ε, ε, εθνικά ομόλογα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αρνητικές αποδόσεις και έχουμε ε, ένα ομόλογο μονοετές, 12 μήνο με συγχωρείτε, με αρνητικό επιτόκιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί που πληρώνει κανείς 3,5% του ΑΕΠ για επιτόκια, που τότε βασικό στόχο είναι να μειωθούν αυτά τα επιτόκια. Όχι μόνο για τη βελτίωση του προπολογισμού, αλλά για να ενισχυθεί η οικονομία. Γιατί έχουμε ένα spillover, γιατί ε, ε, τα επιτόκια για, το εθνικό, για τα εθνικά ομόλογα επηρεάζουν και ε, τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο νοικοκυριών. Πολλέ φορέ όμω έχουμε αναρωτηθεί για, τα αρνητικά επιτόκια ε, ερωτήσει αντιδική σου. Και τώρα η δική σας επιστρέφω στην θέση μου ως ε, Προέδρου του Συμβουλίου και είμαι πεπισμένος πως σήμερα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση παρόλο που υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα τα οποία θίξατε όταν έχει κανείς αρνητικά επιτόκια ε, σε, ένα, σε μια κατηγορία ε, ε, περιουσιακών στοιχείων, τότε ναι μπορεί κανείς να διαφύγει μετακινώντας ε, τις επενδύσεις του ε, σε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Σε εμά, ας πούμε, έχουμε την Αδριατική Ακτή, η οποία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο για μας είναι πάντα προσοδοφόρο και σημαντικό. Οπότε στα πλαίσια του διαλόγου, της δράσης και των στόχων, εμείς ως Προεδρία θα παραμείνουμε στα όσα θα αποφασίσουμε στο Συμβούλιο και στα όσα θα μας πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάριτς. Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις. Θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Παρακαλώ καθίστε, διότι ήδη έχουμε κάποια καθυστέρηση. So, now we are about to start the... Θα ξεκινήσουμε τώρα τη δημόσια ακρόαση με τον προτινόμενο ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών. Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία διορισμού με την οποία ασχολούμαστε σήμερα. Όπως είπα, έχει επιλεγεί ο κύριος Τζέρι Κρός ως νέος εκτελεστικός διευθυντής της CBA. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Κρός η θέση άδειασε στην NBA λόγω της παρέτησης του κυρίου Άνταμ Φάρκα στην 31η Ιανουαρίου του 2020. Η NBA ειδοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Ιανουαρίου του 2020 για την αποφασή της να επιλέξει τον κύριο Κρό σύμφωνα με το ε, ε, ε, δημοσίευμα τύπου της EBA. Τον επέλεξε η EBA από έναν κατάλογο υποψηφίων. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως διευθυντής για τον χρηματοοικονομικό κανονισμό, πολιτική και κίνδυνο στην Κεντρική Τραπεζά της Ιρλανδίας. Η παρούσα δημόσια ακρόαση θα παίξει σημαντικό ρόλο για να υπογραμμίσει τη λογοδοσία του εκτελεστικού διευθυντή της EBA προς το κοινοβούλιο μας. Η ακρόαση βασίζεται στο άρθρο 51 του κανονισμού EBA που προβλέπει ότι ο εκτελεστικό διευθυντή θα διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θητεία είναι πενταετή και μπορεί να παραταθεί μία φορά. Η ακρόση θα έχει ως εξής. Θα έχουμε μια εισαγωγική δήλωση από την υποψήφιο, το πολύ 8 λεπτά και μετά θα εχει ως εξη θα εχουμε μια εισαγωγικη δηλωση απο την υποψηφιο το πολυ 8 λεπτα και μετα θα εχουμε ερωτα απαντησει ε, σε χρόνο 4 λεπτών ένα λεπτό για την ερώτηση και τρία λεπτά για την απάντηση. Θα εφαρμόσουμε τον κανόνα DONT για να καθορίσουμε τη σειρά των ερωτήσεων από τις πολιτικές ομάδες και μετά, αν έχουμε χρόνο, θα έχουμε και catch the eye. Κύριε Κρός, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για αυτή την ακρόαση. Χάρη στι εργασίε αυτή τη Επιτροπή, μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δημιουργήθηκε πριν από 9 χρόνια ω απόκριση στην οικονομική κρίση. Έπαιξε σημαντικό ρόλο για να ε, αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίε τη. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα να λειτουργεί υγιώ, βιώσιμα και δίκαια για να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή οικονομία και εξυπηρετώντα τα συμφέροντα των πολιτών. Για την επιτεύξη αυτών των στόχων η ΕΑΤ απαιτεί σημαντική ηγεσία με στρατηγικό όραμα και οργανωτικές ικανότητες και προσωπικά ε, προσωπικές ιδιότητες κατάλληλες. Υπό την ηγεσία μου η ΕΤΑ θα έχει τις ακόλουθες ικανότητες. Πρώτα απ' όλα κανονισμούς υψηλού επίπεδου μετά από την κρίση θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το κανονιστικό πλαίσιο. Η εκτίμηση αντικτύπου της Συμφωνίας Βασιλείας 3 και οι πολιτικέ συστάσει που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν μια ισχυρή βάση για όλα αυτά. Είναι σημαντικό η ΕΑΤ να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη τη και την επίδραση για να ε, γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε μετά την κρίση. Στο πλαίσιο του Brexit είναι σημαντικό να αποφευθεί οποιοδήποτε κανονιστικό αρμπιτράς που θα υπονόμευε την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό στο έργο αυτό η ΑΕΤ να λειτουργεί ε, στο επίκεντρο. Αυτό είναι σημαντικό για το σωστό κανονιστικό πλαίσιο για να έχουμε ε, πιο απλό πλαίσιο. Σημαντικό εδώ θα είναι η εκπλήρωση της εντολής CRD5 για να γίνει μια ανάλυση των απαιτήσεων με γνώμονα τη μείωση του βάρους για μικρότερες, λιγότερο πολύπλοκες επιχειρήσεις. Ε, Άλλο τομέα προτεραιότητα είναι η υλοποίηση τη αναθεωρημένη τη οδηγία για την εξήγηση των τροπεζών, ούτω ώστε να επανέλθουν οι ευρωπαϊκέ τράπεζε στο επίπεδο που πρέπει και έτσι θα συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Δεύτερον, ενίσχυση τη εμπιστοσύνη και τη αξιοπιστία υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης για να εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας και των ευρωπαίων πολιτών. Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτά τα συμφέροντα. Θα πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργεί δίκαια, ότι λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και ότι επιδιώκει να κάνει αυτό που είναι σωστό και όχι μόνο αυτό που είναι νόμιμο καλύτερη συμπεριφορά, ε, καλύτερη νοοτροπία και προστασία των συμφερόντων και των πολιτών και των τραπεζών όπως και η επίτευξη της πλήρους πολυμορφικότητας σε επίπεδο ε, διευθυντών και ανώτερης διοίκησης. Η εμπιστοσύνη ισχύει και για την ε, ΕΑΤ και η ΕΑΤ θα πρέπει να δρά βάση ποιότητα και εποπτεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν τα μέλη τη λογοδοσία για να παρέχουν υψηλή ποιότητα αποτελεσματική εποπτεία βάσει των αναμενόμενων προτύπων. Επιπλέον θα πρέπει να μάθουμε ε, τα διδάγματα από την, σε διάφορες ε, υποθέσεις Μάρκος Φάρκων. Το σχετικό ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα μας λέει τι πρέπει να κάνουμε συνεργασία, στη συνεργασία της με την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΕΑΤ θα προσπαθήσει να αποφύγει να ξανασυμβεί αυτό. Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά οποιαδήποτε περαιτέρω ε, θέση που μπορεί εγώ να αναλάβω στην ΕΑΤ. Τρίτον, η ε, καταπολέμηση του ξεβλήματος μαύρου χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος. Είναι βασική κίνδυνη για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμείς το λέμε σαφώς ότι οι επόπτες θα πρέπει να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η ΕΑΤ θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για διαμερασμό πληροφοριών για να βελτιώσει την ποιότητα της εποπτείας σε όλες τις δικαιοδοσίες και όπου είναι απαραίτητο για να αξιοποιήσει τις νέες της εξουσίες για να απαιτεί δράση από τις αρμόδιες αρχές. Τέταρτον, βιώσιμη οικονομία. Ο κίνδυνος για το κλίμα και η κλιματική μετάβαση βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή έχουν παίξει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη. Η χρηματοδότηση μια βιώσιμη οικονομία θα αποτελέσει κεντρικό σημείο εστίωση για την επόμενη πενταετία και πέραν αυτή. Ο τραπεζικό τομέα και η ΑΤ θα αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό ταυτόχρονα να μην υπονομεύσουμε το χρηματοπιστωτικό ε, κανονισμό, αλλά ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο έργο τη ΕΑΤ ε, ολόκληρο το πλαίσιο που υπάρχει τριγύρω και τέλος τεχνολογική καινοτομία η οποία μπορεί να φέρει σημαντικά ωφέλη στους καταναλωτές και την οικονομία ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ΕΑΤ στο μέλλον θα είναι ε, η αξιολόγηση ωφελών ε, και κινδύνων ε, με σωστή αξιολόγηση των κινδύνων. Η ΕΑΤ έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα και θα συνεχίσει. Τώρα δύο λόγια για τους μηχανισμούς που θα, για τους κινητήρες δυνάμεις για την επιτυχία στην ΕΑΤ. Η ΕΑΤ απασχολεί 200 περίπου άτομα. Πρέπει να ε, διατηρούν ε, το πνεύμα συνεργασίας ε, κινήτρων και πρέπει να εργάζονται με αξιοπρέπεια, να υπάρχει διαφορετικότητα και να λειτουργούν, πολυμορφικότητα και να λειτουργούν αντικειμενικά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη δική μου εμπειρία στην Κεντρική Τραπεζά της Ιρλανδίας για να αυξήσω την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα τη ΕΑΤ ως οργανισμού. Δεύτερον, οι σχέσεις μεταξύ ενδιαφορομένων είναι κλειδί για την επιτυχία της ΕΑΤ. Η σχέση της ΕΑΤ με αυτήν εδώ την Επιτροπή είχε κάποια προβλήματα και εγώ θα τα διορθώσω. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία και τη διαφάνεια. Ουδέποτε ε, θα ε, παραλείψω τη δέσμευσή μου σε αυτή σε αυτό το επίπεδο. Επίση, ε, όσον αφορά του οικονομικού πόρου, εγώ θα ιδρύσω τη δημοσιονομική πειθαρχία. Βασική ε, πρόκληση θα είναι ο καθορισμό προτεραιοτήτων και η κατάργηση προτεραιοτήτων, ούτω ώστε να χρησιμοποιούμε και του οικονομικού πόρου και τεχνολογία αποτελεσματικά. Και δύο λόγια για μένα. Από το 2015 εγώ υπήρξα μέλο ε, τη ανώτη ηγεσία τη Κεντρική Τράπεζα τη Ιρλανδία, όπου ασχολήθηκα με την χρηματοπιστική πολιτική. Ε, και διεύθυνα 80 και άτομα. Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, ένας οργανισμός υψηλής ποιότητας που βασίζεται στην, ε, στις διαφορετικές ε, ικανότητες του προσωπικού της και που μας καθοδήγησε στο μετασχηματισμό μετά την κρίση. Έχω μεγάλη εμπειρία για να εφαρμόσω ό,τι χρειαστεί προ όφελο τη ευρωπαϊκή οικονομία. Εγώ έχω εργαστεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του Βασιλεία 2. Είμαι μέλο των εποπτών τη ΕΑΤ. Έχω εργαστεί και στον ε, ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Σε όλε μου τι θέσει βασιζόμουν στην πεποίθηση ότι όταν εργάζεται κανεί στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα που επηρεάζει τα δημόσια αγαθά άμεσα. Ω συμμετέχοντε εμεί πρέπει να δράμε με απόλυτη ακαιρεότητα. Αναγνωρίζοντα ότι αν δείξουμε οποιαδήποτε έλλειψη σε αυτό το επίπεδο ή σε άλλα, ζημιώνουμε την ευημερία των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον. Αυτό το πρότυπο υπερασπιζόμουν και είχα θέσει για τον εαυτό μου ανέκαθεν ως εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ πιστεύω ότι θα έχω να αντιμετωπίσω πολλά δύσκολα θέματα και πιστεύω ότι θα μπορέσω να το ε, φέρω εις πέρας επάξια. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στον ε, πρώτο μιλητή Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚΑ για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά, αν μου το επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Καλωσορίσατε εδώ. Έχω δύο σύντομε ερωτήσεις. Πρώτον, τελευταία, διαπιστώνουμε ότι μεταξύ της ΕΑΤ και του SSM ε, υπάρχει κάποιο συναγωνισμός. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός, ποιος είναι ο καλύτερος ε, για την έκδοση εγγράφων και διάφορα τέτοια. Εσείς πώς φαντάζεστε τη συνεργασία με τον SSM, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΑΤ παρά Όλα αυτά θα παραμείνει στην εντολή της. Και η δεύτερη μου ερώτηση για το PSD2 ε, η ΕΑΤ και κατά των τραπεζών και ε, για μας ως ε, καταναλωτές ε, πώς θα διασφαλίσετε στο μέλλον ότι η ΕΑΤ δεν θα καθοδηγείται μόνο από τις τράπεζες, αλλά θα βοηθήσει ώστε στον τομέα της ψηφιοποίησης να αξιοποιηθούν ε, και οι δυνατότητες που προσφέρονται. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Για την ε, σχέση της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Τραπεζών με τον SSM, όταν δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αυτός, και ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα μπρος, μεγάλη σημασίας και πρόκειτο για την ε, ολοκλήρωση της ε, τραπεζικής αγοράς. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ε, και για άλλους. Λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε ο μηχανισμός αυτός, τέθη το θέμα ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ποια είναι σχέση, του της με τον SSM. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν δύο διακριτούς ρόλους και οι οποίοι έχουν λειτουργήσει συμπληρωματικά μέχρι τώρα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Από τη μια, ο SSM έχει αρμοδιότητες για την απευθείας εποπτεία των τραπεζών αυτών, των συστημικών, μέσα στην Τραπεζική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών από την άλλη μεριά έχει θέσει προδιαγραφές για ολόκληρη την ενιαία αγορά και νομίζω ότι αυτό το ρόλο τον έχει παίξει πολύ αποτελεσματικά με τις μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση που είδαμε πως βοήθησαν και άλλαξαν την κατάσταση και σήμερα είμαστε πράγματι σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επικεντρωνόμαστε στην ενιαία αγορά με ενιαίους κανόνες στα πλαίσια του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού, του SSM. Έχουμε συνεισφέρει και εμείς ως ε, ΕΑΤ στην επιτυχία αυτή. Είτε πρόκειται για την βάθυνση ε, και την παγίωση των κανόνων ώστε οι διάφορες ρυθμίσεις να έχουν συνέπεια μεταξύ τους, είτε πρόκειται για τεχνικές προδιαγραφές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχει συμπληρωματικότητα δηλαδή ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και αυτά που κάνει ο νέο εποπτικό μηχανισμό. Τώρα για το δεύτερο, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το δικό μου το πλαίσιο. Οποιοδήποτε σύστημα, μηχανισμό, οργανισμό κτλ. επιδέχεται προκλήσει. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που πιστεύω ότι αξίζουν συζήτηση είναι η προσέγγιση η οποία ε, δημιουργεί ε, πρακτικές και πρότυπα που πρέπει να τηρούνται σε ολόκληρη την έννοια αγορά, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια, όπως είπα, και σωστή εφαρμογή. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, η υγιής ε, συμμετοχή στο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και Ενίου Παπτικού Μηχανισμού είναι κάτι πολύ σημαντικό ήμασταν επιτυχείς μέχρι τώρα. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα δυσκολίες και προκλήσεις, αλλά η σχέση μας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Ρωτάτε τώρα για το PSD και για τον ρόλο Α. Στη Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας εγώ ασχολήθηκα με την καινοτομία και το FinTech. Ένα βασικό στοιχείο εδώ είναι να αντιληφθούμε το φέλη για τα συστήματα και τους καταναλωτές από τις νέες τεχνολογίες, από νέους τρόπους να λειτουργούμε. Και έτσι το σύστημα ανθεί. Δεν λέω να μην σκεφτόμαστε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, φυσικά και πρέπει να σκεφτούμε και να αντιληφθούμε τους κινδύνους που ελοχεύουν, αλλά πρέπει να επιτρέψουμε στην οικονομία να επωφεληθεί από την καινοτομία, τις καινοτόμες ε, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η προσέγγιση να είναι ευρύτερη και τεχνολογικά ουδέτερη. Ευχαριστούμε. Πολ Τάνκ από τους Σοσιαλιστές είναι επόμενος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη προς τον τραπεζικό κλάδο και αυτό νομίζω καλύπτει και τη δική σας στην αρχή και γι' αυτό θα σας ρωτήσω για την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Ως, ως, ε, ως μέλος λοιπόν εσείς ε, του Διοικητικού Συμβουλίου που υποπτεύει ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή. Εσείς ε, ήσασταν, ε, παρακολουθήσατε τη μεταφορά του κυρίου Φάρκας στην άλλη υπηρεσία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι έγινε, πώς αντιμετωπίζετε τα θέματα του τραπεζικού λόμπινγκ δεδομένης και της υπόθεσης αυτή. Και δεύτερον, ε, μόνο μία γυναίκα έχετε στο δικαιωτικό συμβούλιο. Μόνο μία γυναίκα είναι στο εποπτικό σας συμβούλιο. Συμφωνείτε με την αρχή πως για κάθε θέση θα πρέπει να έχετε υποψηφιότητα και γυναικεία και ανδρική ε, που θα ε, στέλνετε στο κοινοβούλιο για να λάβουμε εμείς την απόφαση. Και για να έχουμε ισότητα μεταξύ των φίλων στην λήψη οικονομικών αποφάσεων, τι ε, σκοπεύετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπόθεση Φάρκα, στην οποία περιέγραψα να σας πω πως Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντικό και θεωρώ ότι θα μετατρέψει ε, την ε, κατάσταση και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ε, παρακολουθούμε τέτοιες υποθέσεις και τις διαχειριζόμαστε. Όταν κάποιο δηλαδή φεύγει από μια εξαιρετικά υψηλή θέση από το δημόσιο και μεταφέρεται στον ιδιωτικό κλάδο, πρέπει να γνωρίζουμε, ε, να ε, δούμε τι θα κάνει με τι γνώσει που έχει αποκτήσει εκ των έσω και πώ θα τι χρησιμοποιήσουν ή όχι. Δεύτερον, το γεγονός πως ενδεχομένως επηρεάζουν ε, αυτούς τους οποίου έχουν εργαστεί για του ίδιου ή για του οποίου οι ίδιοι έχουν εργαστεί. Και τρίτον, τα κίνητρα στο σύστημα στην περίπτωση όπου υπάρχει εύκολη μετάβαση από υψηλά ιστάμενη θέση στο δημόσιο κλάδο προς τον ιδιωτικό. Αυτό ε, δυστυχώς ε, ε, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ε, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο κλάδο αντιμετωπίζουν τις δυνατότητες καριέρας και ανέλυξης στον ιδιωτικό. Ε, και αυτό δημιουργεί ε, αθέμητες καταστάσεις. Τώρα, για το θέμα της επιβολής και τα όσα είπατε, ναι, πολύ σωστά το έχετε φωτίσει και θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε αν μπορούμε πραγματικά να βρούμε τρόπους για να επιβάλλουμε τις αποφάσεις μας αλλά γενικότερα το γεγονός πως υπάρχει ε, ανάγκη μιας περίοδος cooling off, δηλαδή ενός διαστήματος κατά το οποίο δεν επιτρέπεται αυτή η μετάβαση, μπορούμε να το εξερευνήσουμε, να έχουμε κάποιες επιπλέον δεσμεύσεις, αλλά να το κάνουμε σαφές. Εάν έχεις υψηλή θέση στο δημόσιο κλάδο και θες να μετακινηθείς στον ιδιωτικό κλάδο, και νομίζω ότι εδώ είναι καλό το παράδειγμα, τότε θα πρέπει να ε, υπάρχει μια περίοδος όπου μπαίνει στο ψυγείο κατά κάποιο τρόπο. Και μπορώ να ε, δεσμευτώ πως θα έχουμε τέτοιου είδους, αν θέλετε στην περίπτωσή μου, διετή ε, περίοδο μη μετακίνησης. Νομίζω ότι χρειάζεται μία επίγουσα τροποποίηση και αυτό να το τοποθετήσουμε και στο πλαίσιο του ε, ε, καταστατικού μας τώρα για το ρόλο μεταξύ ε, της δικής μας αρχής και της ΑΦΜΙΤ να σας πω πως στα πλαίσια της προσπάθειας μετά την κρίση να επανειδρύσουμε το σύστημα παρακολούθησης θεωρούσα πως το πιο σημαντικό ήταν ο κλάδος να δει πως συνομιλεί με τον νομοθέτη. Γιατί είχαμε βρει ένα βαθμό ε, συγχώνευσης μεταξύ ε, βιομηχανίας και ε, εποπτικών και κανονιστικών αρχών που ήταν ενδεχομένως υπερβολικός όπου ε, τα συμφέροντα της βιομηχανίας θεωρείται ότι ταυτίζονται με τα δημόσια συμφέροντα και αυτό μετά την κρίση κατέρευσε ως ε, σχήμα και έβλαψε πάρα πολλούς πολίτες ακόμα και στη δική μου χώρα. Μετά την κρίση λοιπόν χρειάστηκε να αλλάξει ο κλάδος τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ε, με τον νομοθέτη και χρειαστήκαμε να βρούμε τα κατάλληλα άτομα. Εγώ ανέλαβα το ρόλο λοιπόν και στις δύο αρχές, λέγοντας πως εάν επιθυμούμε να αλλάξουμε θα χρειαστεί να βρούμε άτομα τα οποία ε, θα ε, ε, παρέμβουν έτσι ώστε η, η βιομηχανία, ο κλάδος ολόκληρος να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι η δική μας στάση είναι πολύ σημαντική. Είμαστε οι αρχές οι οποίες εξασφαλίζουν πως η συμπεριφορά ε, των ε, εμπλεκομένων είναι η σωστή και θα πρέπει όσοι εργάζονται στις δύο αρχές να έχουν μια στάση η οποία είναι αναλογική, είναι ανεξάρτητη, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία, ε, συνετή έτσι ώστε να μπορούμε στις πληροφορίες που λαμβάνουμε να μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή stop μέχρι εδώ. Για το θέμα της διαφορετικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην ε, Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας το έχουμε ε, ως κεντρικό ε, αναπόσπαστο σημείο. Εγώ στο κλάδο μου έχω μονάδες στις οποίες είμαστε 60% γυναίκες, 40% άνδρες, οπότε πιστεύω πως χρειαζόμαστε τη διαφορετικότητα, όχι μόνο δηλαδή διαφορετικά φύλλα, αλλά όλων των ειδών τις διαφορετικές προελεύσεις και ομάδες. Η Στεφανή τη Ρημνιού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτές που έκανε και ο συνάδελφος Πολτάγκη. Η πρώτη σχετίζεται με το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που η Επιτροπή μας θέλει να καταπολεμήσει ε, απόλυτα. Την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ενός ψηφίσματος ΕΚΟΝ που καλεί τα διοικητικά συμβούλια ε, της ε, ΕΑΤ που επέτρεψε στον κύριο Φαρκάς να εργαστεί εκεί σε αυτή τη θέση που ανέλαβε μετά από τη θέση που κατήχε. Η δική σας κατάσταση είναι η ίδια, αλλά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει και εσάς, γιατί και εσείς ε, ήσασταν διευθυντής εκεί για τέσσερα χρόνια πριν τώρα σας διορίσουν ως υποψήφιο. Αυτό το ψήφισμα της περασμένης Πέμπτη υπογραμμίζει αυτό το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται, όπω είπα, με το σύστημα αυτό που υπάρχει περίπτωση να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη ε, στους θεσμικά όργανα των πολιτών μας. Ε, ξέρετε, η αξιοπιστία του θεσμού είναι ύψη της προτεραιότητας. Πώς λοιπόν στη δική σας περίπτωση θα απομακρύνετε οποιαδήποτε υποψία σύγκρουση συμφερόντος και θα αναλάβετε με απόλυτη αυτονομία και αμεροληψία τη θέση σας. Η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με μία από τις ε, προτεραιότητες ε, υπέρ ε, της καλύτερης ανάμειξης για να μην πω ισοδυναμίας γυναικών και ανδρών στην Νέα Θητεία. Αναρωτιέμαι τώρα, αντί για μια δέσμευση, θα με μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει εδώ στην ΕΚΟΝ, δεν υπήρξε καμία γυναίκα υποψήφιος με αντίστοιχα φυσικά προσόντα για ακρόαση. Εσείς ως εκτελεστικός διευθυντής τι θα κάνετε διότι δεν άκουσα να λέτε κάτι για συγκεκριμένη δράση ώστε να διασφαλίσετε αυτή την πολυμορφία εντός της ΕΑΤ. Αυτά. Thank you for that. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που κάνατε για το πώς εγώ θα διασφαλίσω την αξιοπιστία της ΑΦΜΗ και την αποφυγή να, τη σύγκρουση συμφερόντων. Να σας πω το εξής πολύ σαφώς. Εργαστικά για πέντε χρόνια. Έχουν περάσει μάλλον πέντε χρόνια από τότε που εργαζόμουν στην ΑΦΜΕ. Όπως ανέφερα αυτό το ζήτημα των ανθρώπων που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και μετά ε, στον ε, κρατικό και το αντίστροφο. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Transparency International μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχει ε, αναφέρει και τις αρχές ε, απασχόληση ανθρώπων στον ιδιωτικό τομέα και μετά στον κρατικό ε, ή πρώτα στον κρατικό και μετά στον ιδιωτικό έχει κάποια ωφέλη εφόσον γίνεται σωστά. Δεν λέω εγώ ποιε πρέπει να είναι περίοδε, δεν λένε ποιε περίοδοι πρέπει να υπάρχουν. Λένε ότι αυτή η περίοδο αναμονή ενό-δύο έτων είναι εντάξει. Έχουν περάσει πέντε έτη από τότε που εργαζόμουν εγώ στην ΑΦΜΗ και πιστεύω ότι αυτό το διάστημα απομακρύνει οποιαδήποτε αίσθηση ότι έχω και στενές επαφές με αυτόν τον οργανισμό στον οποίο ναι μεν εργάστηκα στο παρελθόν. Δεύτερον, στο διάστημα αυτό εγώ δραστηριοποιήθηκα στο... και πρόθεσα κανονιστικές προσεγγίσεις και αλλαγές που σίγουρα δεν ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα κάποιων βιομηχανιών. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία, το τελευταίο καιρό όπως τα γνωρίζετε, είχαμε να κάνουμε με το Brexit και το τι θα σήμαινε το Brexit για τις Ιρλανδικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Υπήρξε τεράστια πίεση από διάφορους ε, φορείς που μας έλεγαν, από διάφορους ενδιαφερομένους που μας έλεγαν ότι δεδομένου ότι όλες αυτές οι εταιρείε πρέπει να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα ήταν καλό να έρχονταν στην τάδε δικαιοδοσία ή στην δίνα δικαιοδοσία. Δεν θα ήταν καλό να ε, τις... Ε, βολέψουμε κάπως με κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση. Εμεί στην Ιρλανδία είπαμε πολύ καθαρά ότι δεν θα συμβιβαστούμε όσον αφορά τα πρότυπά μα ότι δεν θα προσπαθήσουμε ω ρυθμιστική αρχή να προωθήσουμε ή να προσελκύσουμε κάποιες τράπεζες σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίε. Κάναμε, ακολουθήσαμε μια πολύ διαφανή γραμμή. Είπαμε ότι αν θέλουν να εγκατασταθούν στην Ιρλανδία ε, τράπεζες πρέπει να έχουν ουσιαστική παρουσία στη δικαιοδοσία μας και να πληρούν όλες τις απαιτήσει και τα πρότυπά μας χωρίς καμία προσαρμογή ή υποχώρηση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ήθελα να σα αναφέρω τι κάνω αυτή τη στιγμή. Ε, διευθύνω την υλοποίηση ενός πλαισίου ε, ατομικής λογοδοσία για τι χρηματοπιστωτικές μα εταιρείε. Και ένα από τα πράγματα που έχω αναφέρει είναι ότι είναι σημαντικό να αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά. Στην Ιρλανδία είμαστε μία από τι ελάχιστε χώρε στην Ευρώπη που κανονιστικά προσπαθούμε να εισάγουμε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου τα ανώτατα διοικητικά στελέχη θα απαιτείται να λένε ρητά για ποιο πράγμα είναι αρμόδιοι σε πλαίσιο ποια δομή μέσα σε έναν οργανισμό και πώ ε, πληρούν τα πρότυπα, τα σαφή πρότυπα και να, είναι, να λογοδοτούν για αυτά. Οπότε Πιο συγκεκριμένα, αν μου επιτρέψετε για το ζήτημα τώρα της ε, ε πολυμορφίας. Για να απαντήσω στον κύριο Τάγκ, είναι πολύ σημαντικό ε, και αυτό το μάθημα από την κρίση. Να σκεφτώ... Ε, η ομαδική σκέψη είναι αυτή που μας οδηγεί σε δυσκολίες. Σε ό,τι κάνω, για μένα είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ε, ισορροπία και στη διάσταση του φύλου και με άλλου τρόπου όσον αφορά του υποψηφίου, και αυτό έχω επιτύχει και εγώ στη δική μου διεύθυνση στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Το τι γίνεται στην ΕΑΤ και από ό,τι κατάλαβα υπήρχε μία. Ε, στο, κατάλογο, στο τελικό κατάλογο υπήρχε και μια γυναίκα ε, υποψήφια. η διαφορετικότητα την υπερασπίζονται αρκετά έντονα στην ΕΑΤ και θα διατηρηθεί έτσι. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μία ερώτηση παρακαλώ και ένα λεπτό για αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε όλε τις απαντήσεις. Σβέν Γκίγκολτ, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Τονίζω ότι για μένα εδώ δεν μιλάμε για ένα κλασικό θέμα cooling off, δηλαδή περίοδου ανάμεσα στις ε, δύο θέσεις. Το θέμα που πρέπει εδώ να απαντήσουμε είναι κατά πόσο σε αυτή την κατάσταση είσαστε ο κατάλληλος για να βρεθείτε επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και εδώ θα ήθελα σαφή απάντηση στην ερώτηση του συναδέρφου Τάγκ, που είναι τι ρόλο παίξατε στην απόφαση για τον κύριο Φάρκας. Δηλαδή εσείς στο Συμβούλιο Εποπτών τι θέση πήρατε, ζητήσατε μεγαλύτερη περίοδο cooling off δεσμευτικά. Δεύτερον, για οποιοδήποτε μέλος του Ποπτικού Συμβουλίου, όταν αποφάσισε για την Dansk Bank, εσείς τι ψηφίσατε, πώς τοποθετηθήκατε για να προστατεύσετε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Αυτές είναι οι δύο μου ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. για να απαντήσω στην ε, πρώτη ερώτηση. Όπως είπα, όταν δούμε το καταστατικό και το έργο της Επιτροπής σας αυτής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αλλάξει. Τώρα είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που είμαστε νωρίτερα. Αν δείτε λοιπόν το κείμενο του εσωτερικού κανονισμού που διέπει αυτά τα ζητήματα, στην διατύπωση, στην διάρθρωση των περιορισμών και των δικαιωμάτων προκειμένου να μπορεί να κερδίζει κανείς ε, το ψωμί του, πολύ συχνά μιλάμε για τη σύγκρουση συμφερόντων και πώς αυτή αντιμετωπίζεται μέσω αυτών των περιορισμών ακριβώς αν δούμε το κείμενο που έχει οθετήσει η Επιτροπή, είναι αυτό το κλασικό που εγκρίνεται. Τώρα εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αλλάξει. Όσον αφορά γιατί με ρωτήσατε. Εγώ ζήτησα να σκληρύνουν οι όροι. Αλλά δεν είπα ότι πρέπει να υπάρξει απαγόρευση. Αν ξαναβρισκόμασταν μπροστά στην ίδια περίπτωση, πολύ πιθανόν να έλεγαν «Ναι, ναι, υπάρχει απαγόρευση. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν όμως ήταν απόφαση της ΕΑΤΕ, λέει ο κ. Γκίγκολτ. Όχι. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας. Τράπεζα Ντάνσκ. Εδώ υπήρξε μια παραβίαση της νομοθεσίας ε, όσον αφορά τη Δανία και την Εστονία. Η δικιά μου άποψη ήταν και είναι ότι υπήρχε πρίμα φάτσε απόδειξη, υπήρξαν μαρτυρίες για λάθη και αδυναμίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν μια περίπλοκη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα είχαμε να κάνουμε με δραστηριότητες που συνηθίζονταν στο παρελθόν, με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο άλλαξε στο μεταξύ και υπήρχε το ζήτημα και παραμένει σε τι βαθμό οι εποπτικές αδυναμίες αποτελούν παραβίαση της νομοθεσίας. Εγώ έλεγα ότι πολύ πιθανό ναι, να υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Και αυτό το οποίο είπα στο Εποπτικό Συμβούλιο ήταν ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία. Ότι χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο να διερευνήσουμε την υπόθεση. Η απόφαση όμω ήταν ότι περιοριζόμασταν από τους δύο μήνες που προβλέπει η νομοθεσία και δεν είχαμε παραπάνω χρόνο. Τώρα εφ' εξή, θα έλεγα ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό το στοιχείο, γιατί πράγματι ε, θα πρέπει να μπορούμε να διερευνήσουμε αρκετά για να ε, λογοδοτούμε. Εσείς καλύπτετε την ε, απόφαση, δηλαδή εσείς υπερψηφίσατε την απόφαση να μην ε, υπάρξει παρετέρω διερεύνηση. Όχι. Η θέση μου ήταν ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Μα τι ψηφίσατε, υπέρ ή κατά. Μα τότε τα ε, στοιχεία δεν μπόρεσαν να διαρρευθούν αρκετά γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Ωραία. Ε, ID τώρα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω γερμανικά και έχω δύο ερωτήσεις. Θα ρωτήσω την πρώτη και αν έχω χρόνο θα κάνω και τη δεύτερη. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση κινδύνου, στατιστικά για το τρίτο τρίμηνο του 2018 τα κέρδη από μετοχές τα 7 από τα 9 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν. Ε, στα υπόλοιπα μειώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησαν πως εδώ έχουμε αρνητικό, αρνητικό αντίκτυπο. Οπότε εσείς πώς αντιμετωπίζετε τη χαλαρή νομισματική πολιτική ε, της ε, ΕΚΤ για το θέμα αυτό ε, και κυρίως για τις τράπεζες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε μια συγκυρία που δεν τρέχει με τη μέγιστη ταχύτητα. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές προκλήσεις. Τα αρνητικά επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια είναι προβληματικά ε, ως περιβάλλον, όχι για μένα, ε, βέβαια δεν είναι για μένα να πω το ποια θα έπρεπε να είναι, γιατί εγώ απλώς είμαι επόπτης, αλλά θα πρέπει να δούμε την όλη διάσταση του ζητήματος και ένα από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι η μείωση της ε, κατάτμισης στην ενιαία αγορά και στην Τραπεζική Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες μετά την κρίση έχουν κλειστεί μέσα στα εθνικά του σύνορα και παίζουν όλα ένα παιχνίδι αναμονής μέσα σε ένα περιορισμένο ε, περιβάλλον ε, αγορά, οπότε θέλουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, λιγότερη κατάτμιση και μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο άνοιγμα σε άλλες αγορές. Τα επίπεδα του λόγου κόστους εσόδων των τραπεζών δεν έχουν μειωθεί με τον τρόπο που ε, θα ήθελα να έχω δει, έτσι ώστε να έχουμε ε, καλύτερη απόδοση και μείωση του κόστους, αλλά ένα κομμάτι του ρόλου μας ως εποπτικό όργανο είναι να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια ε, και να κάνουμε την αξιολόγηση κινδύνου στην οποία εσείς αναφερθήκατε και να την, και... να τη διανύμουμε. αυτή τη στιγμή οι τράπεζες λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, έχουν ε, μικρότερη ε, αξία από ό,τι είναι εγγεγραμμένοι στα περιουσιακά τους στοιχεία και νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να παρουσιάζουμε αυτές τις πληροφορίες, να τις ερμηνεύουμε, να μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει, να κάνουμε τα stress test, να κάνουμε την αξιολόγηση κινδύνου και αυτή τη στιγμή νομίζω εκεί βρισκόμαστε γιατί τρέχει μια διαβούλευση για ένα θέμα που είναι τι μορφή θα πρέπει να έχει το επόμενο stress test για τις τράπεζες. Τεστ ανθεκτικότητας δηλαδή. Τώρα τα χαμηλά και αρνητικά επιτόκια είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τράπεζες και εμείς έχουμε ως ρόλο να εξασφαλίσουμε ότι ο κλάδος θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά α, σωστά. Από την ECR, ο Eugene Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα του μηδενικού κινδύνου για τα ομόλογα. Ποια είναι η δικιά σας θέση για την σχέση των τραπεζών με τα κρατικά ομόλογα και την διάσωση των τραπεζών. Ευχαριστώ. Μετά την κρίση, την ε, κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, φάνηκε ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, η σχέση τραπεζών ε, με δημόσιο χρέος και την εξάρτησή τους από το δημόσιο χρέος, φάνηκε πόσο σημαντικό ήταν. Και οι νομοθέτες και εμείς κάναμε πρόοδο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά εργαλεία τα οποία βοηθούν Βέβαια το βασικό είναι η οδηγία για την ανάκαμψη και την ε, εξυγένση των τραπεζών. Τώρα πια στην νομοθεσία υπάρχει η άποψη ότι όταν ε, είναι σε πρόβλημα οι τράπεζες είναι οι μέτοχοι που αναλαμβάνουν το ρίσκο δεν έχουμε φτάσει ακόμα ώστε σε σημείο που να λειτουργεί πλήρως και επιτυχώς το σύστημα. Υπάρχει η δεύτερη οδηγία BRDT που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε περισσότερο. Τώρα περνάμε στο θέμα της ε, εξυγίανσης η καθάριση των τραπεζών. Έχουμε τον πυλώνα 2 και 3 της Τραπεζικής Ένωσης ώστε να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει η ρευστοποίηση, ότι μπορεί να υπάρξει προστασία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πάντως, κάτι σημαντικό είναι το πώς χειριζόμαστε το θέμα του μηδενικού ρίσκου από τα κρατικά ομόλογα. Οι αρμόδιοι είπαν ότι δεν θα πρέπει απόλυτα να υπάρχει μηδενικό ο κίνδυνο για τι διάφορε μορφέ, πάντω δεν είναι οι ρυθμιστέ που αποφασίζουν. Είναι ένα νομοθετικό ζήτημα το οποίο πρέπει οι νομοθέτες να χειριστούν. Ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις για το πώς μπορεί να γίνει με συγκέντρωση και δίνουμε άλλα μέσα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται σε επίπεδο ένα. Πάντως από τη δικιά μας την πλευρά είναι σωστό να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση του κινδύνου. Ωραία. Χωσέ Γκουσμάλα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως η αξιοπιστία ε, της αρχής σας ε, έχει πληγεί πάρα πολύ από την υπόθεση Φάρκας και ενώ αληθεύει πως οι κανονισμοί του επέτρεπαν και το καταστατικό, πρέπει να δούμε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση, γιατί θα έπρεπε να έχετε προστατεύσει ε, την ε, κοινή γνώμη, γιατί όταν ένα λόμπι έρχεται και ψάχνει έναν ένα νομοθέτη σε υψηλή θέση ε, σε έναν οργανισμό, τα πράγματα δεν είναι καλά. Αυτό συνέβη με την υπόθεση Φάρκας και οι περιορισμοί που είχατε θέσει ήταν γελίες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως η πρόταση διορισμού σας ε, δείχνει πως έχει μια έλλειψη ευαισθησίας η αρχή σας. Το ψήφισμα βέβαια που εμείς δημοσιεύσαμε δεν χρησιμοποιήθηκε όσο θέλαμε, γιατί δεν περνάει κανείς από ένα δημόσιο, μια δημόσια θέση σε μια ιδιωτική ε, με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι απολύτως νόμιμη, που να μην δημιουργεί πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι φεύγουμε από μια υψηλά θέση, στο, υψηλή θέση στο δημόσιο και αυτός ο οποίος δημιουργεί τους κανόνες μένει στον ίδιο κλάδο και κάνει lobbying σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Ε, αυτό δεν θα έπρεπε να το επιτρέπετε και νομίζω πως και ο πρόεδρος της αρχής σας δεν θα έπρεπε να το επιτρέπει και δεν θα έπρεπε ε, να, το, να έχει γίνει στην υπόθεση φάρκα αυτό ζεστό, ε, δεκτό και επίσης με το διορισμό που συζητάμε σήμερα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Χρειάζεται να κάνουμε καλύτερες επιλογές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε κάτι το ίδιο ε, στο μέλλον. Σας, ε, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις διευκρινήσεις σας, αλλά ακόμα δεν μας έχετε πει. Τι θα κάνετε Πώς θα εξασφαλίσετε την ισορροπία ε, μεταξύ των δύο φύλων, αν εσείς ε, διοριστείτε σε αυτή τη θέση. Θέλω να ξαναπώ για το θέμα αυτό του κυρίου Φάρκας και της ΑΦΜΗ, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό μετά, μετά την κρίση ο κλάδος να αλλάξει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται. Ήταν πολύ σημαντικό να σταματήσει να έχει τις στενές σχέσεις και να κάνει το lobbying που γινόταν πριν την κρίση και να πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ο κόσμος χρειαζόταν να αναλάβει τις ευθύνες για τα όσα είχε κάνει. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη μου. Ανέλαβα το ρόλο αυτό και πιστεύω πως έκανα πολύ καλή δουλειά. Και είπα έτσι από εδώ και πέρα θα προσεγγίζουμε, Βασιζόμαστε στα πιστήρια και στα δεδομένα. Είμαστε ήρεμοι και προσεγγίζουμε τα θέματα για να δώσουμε μια καλή λύση. Εγώ, ε, για παράδειγμα, δεν είχα ποτέ κάρτα για να μπαίνω στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί? Γιατί εγώ έπρεπε να κάνω την έρευνα, να σας στείλω τα δεδομένα, να σας στείλω ε, τα πιστήρια. Αυτό και τι αποδείξεις. Αυτό χρειαζόμαστε από όλου για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Πιστεύω πω τα καταφέραμε. Τώρα, είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί ότι παρόλο που δεν έχετε παίξει αυτό το ρόλο για πέντε χρόνια, θεωρούμε πως και πάλι δεν είναι σωστό. Το κάνατε για τους κατάλληλους λόγους, ήσασταν πετυχημένους, πετύχατε αυτά που θέλατε, είστε εκτός ρόλου για πέντε χρόνια, αλλά παρόλα αυτά μας δεν μας αρέσει. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Και για την ισορροπία μεταξύ ισορροπή, ε, εκπροσώπηση των δύο φύλων πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό. Εκεί που εργάζομαι τώρα, για παράδειγμα, έχουμε πολύ ευέλικτες συνθήκες εργασίας, είναι πολύ φιλικό προς τις οικογένειες στο περιβάλλον, Έχουμε μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση στις γονικές άδειες, στην εργασία από το σπίτι, στη, ε, ε, μειωμένο ωράριο αλλά βέβαια πρέπει να προωθούμε και τις κατάλληλες αιτήσει. Οπότε θεωρούμε ότι στη δική μας τράπεζα ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως ε, άνθρωποι που έχουν φύγει με ε, γονική άδεια ε, επανέρχονται γιατί έχουν τις δεξιότητες τους, έχουν τις ευθύνες τους, έχουν το τι έχουν μάθει μέχρι σήμερα και μπορούν να συνεισφέρουν και έτσι. Και βέβαια θέλει κανείς να εξασφαλίσει πως ο κατάλογος των όσων υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης επιτρέπει κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να είμαστε φιλικοί προς αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει κάποιο χρόνο εκτός και θέλουν να επιστρέψουν. Μπορούμε να κάνουμε πολλά λοιπόν. Γιατί θέλουμε να έχουμε ένα περιβάλλον εργασιακό στο οποίο εκπροσωπούνται ισότιμα τα δύο φύλλα. Ευχαριστούμε. Έχουμε καθυστερήσει. Ε, θα καθυστερήσουμε για 10 λεπτά, αλλά πολλοί κόσμος έχει ζητήσει το λόγο για το Catch the Eye. Ήθελα να δώσω λίγο χρόνο γι' αυτό, αλλά να είστε πολύ σύντομοι και πολύ ακριβείς. Και υπό την προπόθεση ότι θα περικόψουμε λίγο από το επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξη. Ε, μόνο έτσι. Ούτως ή άλλω θα ψηφίσουμε αύριο. Οπότε να συναντηθούμε. γι' αυτό. Συμφωνούμε επί αυτού Ωραία, πάμε λοιπόν στο πρώτο κατσδία. Ένα λεπτό, ήταν Χούμπνερ, ΕΛΠΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα ρωτήσω όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης του κινδύνου και των δικτών διαμερισμού του, καταμερισμού του κινδύνου. Τι μπορεί να κάνει η ΆΤΑ για αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. So, so I think Πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πολύ αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση του RRG2 που ψηφίστηκε εδώ πρόσφατα. Είναι πολύ σημαντικό όπως ανέφερα να επιτευχθεί η ρευστότητα των τραπεζών, να επιτυγχάνεται όσον αφορά ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPL που είναι βασικός δείκτης, ε, το ξέρω και εγώ από τη δική μου δικαιοδοσία, το γνωρίζω ε, από πρώτο χέρι, είναι το πόσο σημαντικό είναι να μειωθούν ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπερασπίζουμε το συμφέρον των ανθρώπων που έχουν λάβει δάνεια και των καταναλωτών. Ε, κάτι επιτυχημένο που κάναμε στην Ιρλανδία ήταν ότι δημιουργήσαμε ένα κώδικα διοντολογίας για τα ενυπόθηκα αυτά δάνεια, ούτω ώστε και για τις καθυστερούμενες πληρωμές ε, και με αυτό μπορεί κανείς να καθορίσει μετά διευθετήσεις για το πώς θα χειρίζονται οι τράπεζες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτείται εποπτική παρέμβαση, απαιτείται από τις τράπεζες ε, για κάτι τέτοιο να έχουν τις δομές, τους εμπειρογνώμονες, ε, τη βούληση, να ασχοληθούν με αυτά, πρέπει να έχουν σαφείς στόχους, ε, να είναι διορατικές, δεν υπάρχει τέλεια λύση. Υπάρχουν και διάφορες άλλες λύσεις που επινοήσαμε και η ΕΑΤ βρήκε μια πολύ καλή λύση. Ανέπτυξε κριτήρια για την τιτλοποίηση και διασφάλισε να χρησιμοποιηθούν διάφορες μεθοδολογίες και φυσικά κάτι σημαντικό που έκανε η ΆΤ είναι ότι ε, δημιούργησε ορισμούς και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αυτό μας βοήθησε να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Για να επιταχύνουμε τη διαδικασία θα κάνουμε το εξή. Τρει ερωτήσει μαζεμένες και η απάντηση θα είναι και για τις τρεις. Παρακαλώ. Εσείς, κύριε Γκόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τις απαντήσεις σας και για την ισότητα των φίλων, την ισορροπία μεταξύ των δύο και τις άλλες απαντήσεις που μας δώσετε. Είναι καλό να δίνετε ευκαιρίες στις γυναίκες και χαίρομαι που το Συμβούλιο Εποπτών στην ΕΑΤ έκανε σύσταση για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για την ε, θέση. Και βλέπω ότι σας ρωτούν από τη δεξιά για την ουσία, ενώ σας ρωτούν για τους τύπους από την αριστερά. Ποια είναι η ερώτησή μου. Ωραία, είναι για τις χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μια νέα προϋπόθεση για τις χώρες αυτές, πώς θα ενταχθούν στο ευρώ και στην Τραπεζική Ένωση. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την προϋπόθεση λειτουργεί και ποια είναι η εμπειρία που έχετε όντας επόπτης για την προετοιμασία που κάνουν οι χώρες αυτές. Ρόμπερτ Ρόλεντ, μη εγγεγραμμένος. 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση, παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι κατά πόσο πιστεύετε από τη δικιά σας χώρα, την Ιρλανδία, ε, με τα αρνητικά ή πολύ χαμηλά ε, επίπεδα επιτοκίων, πώς ε, επηρεάζει αυτό τα ενυπόθηκα δάνεια ο δανεισμό μάλλον προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν αυξάνεται. Μήπως αυτό θα μας οδηγήσει σε μια νέα φούσκα που θα ξεσπάσει στα μούτρα μα αργότερα. Ευχαριστούμε. Τελευταίος, Φράσις Φιτζέραλτ. Έλκ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε πως τα τελευταία πέντε χρόνια ρυθμίζεται το Ιρλανδέζικο τραπεζικό σύστημα σε μια εποχή μετά την κρίση με ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω Brexit. Ξέρω τι έχετε κάνει για την ισότητα των φύλων, την ακυριότητα την προσωπική σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για την ηθική διοντολογική συμπεριφορά στο τραπεζικό σύστημα. Τι μπορείτε να αλλάξετε, δεδομένων των όσων έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και δεύτερον, ποια είναι τα διδάγματα από την Ιρλανδία και από τι εμπειρίε που έχετε αποκτήσει για την εποχή ε, για την εποχή ε, την επόμενη και για, μετά τα όσα συνέβησαν στην αρχή σας. Έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε. Thank you. Um, I Για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, να σας πω πως πάντα ήταν ανοιχτή στα μέλη εκτός ευρώ, αλλά η λογική είναι αν έχεις κοινό νόμισμα, τότε να έχεις και μια κοινή προσέγγιση, ενιαία προσέγγιση στον τρόπο που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σου σύστημα. Ενιαίο υπόπτη, για παράδειγμα, ε, ένα ε, ενιαίο μηχανισμό επίλυσης ε, και ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Χωρίς αυτά, τι συμβαίνει. αυτός ο κύκλος, ε, ο επικίνδυνος ε, με επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν και επανέρχονται κυκλικά. Γιατί οι εθνικές τράπεζες αποκτούν μια περίεργη σχέση με, τις, ε, το κράτος τους από τη στιγμή που ανήκουν επίσης και σε ένα ευρωπαϊκό νόμισμα. Οπότε Τραπεζική Ένωση είναι σημαντική, δημιουργεί θέματα, κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν. Οπότε, κανονιστικά ομιλώντας ε, και όχι πολιτικά, Πιστεύω πως υπάρχουν τεράστιες συνέργειες και πλεονεκτήμα από το να έχει κανείς έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που όλοι ως κοινότητα εποπτικών αρχών συνεργαζόμαστε σε μεικτά κλιμάκια, ε, μοιραζόμενοι τις εμπειρίες μας και τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν. Σε αυτά είναι καλύτερη η Ευρώπη. Οπότε, ναι, τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Και στη δική μου χώρα έχουμε υποφεληθεί. Για τα αρνητικά επιτόκια και για το περιβάλλον που δημιουργούν εγώ δεν μπορώ να τα σχολιάσω, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Δημιουργεί πολύ συγκεκριμένες συγκυρίες οι οποίες διαμορφώνουν το πώς αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που αναδύονται ή όχι. Άρα λοιπόν ε, αγορά κινήτων και άλλα είδη περιουσιακών ε, στοιχείων όπου μετακινούνται εκεί οι επενδύσεις και ενδεχομένως δημιουργούν φούσκες με τα γνωστά προβλήματα επίσης. Το θέμα του μη τραπεζικού ε, κλάδου. Και εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος ε, φούσκας. Οπότε ναι, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι αυτοί όταν μιλάμε για άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός τραπεζικών ε, Και αυτά πάντα υπό το φως των διδαγμάτων που λάβαμε από την προηγούμενη κρίση. Για το ηθικό θέμα που θέσατε είναι τεράστιο και στην Ιρλανδία και όλοι μας και εγώ προσωπικά εστιάζουμε ιδιαίτερα στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί με έναν τρόπο όπου οι άνθρωποι πραγματικά εμπιστεύονται το σύστημα αυτό. Ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει και για να το πετύχουμε χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία μας οι τράπεζε θα πρέπει να αναρωτιούνται όχι μόνο μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά θα έπρεπε να το κάνω αυτό, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα από τους βασικούς μηχανισμούς τους οποίους εμείς επιδιώκουμε και η κυβέρνησή μου προσπαθεί να νομοθετήσει έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο ξεκάθαρο για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις ε, ε, όσων βρίσκονται σε υψηλές θέσεις management πώς δηλαδή αυτοί οι υψηλά ιστάμενοι μάνατζερ πρέπει να συμπεριφέρονται με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα τους επιτρέπει να επιβάλλουν αυτή την ηθική. Τέλος, διδάγματα από την Ιρλανδία. Πολλά και οδυνηρά. Και θα έλεγα πως γνωρίζουμε ποια είναι η σημασία αν είσαι ρυθμιστής να γνωρίζεις τι προσπαθείς να πετύχεις. Είσαι υπεύθυνος για να εξασφαλίσεις τη χρηστότητα, την ασφάλεια, την ορθή συμπεριφορά του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού κλάδου. Αυτά μόνο. Οτιδήποτε που τα υποσκάπτει θα πρέπει να αποφεύγεται και αυτά θα πρέπει να διαφυλάξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρός. Ας α, περιμένουμε ένα λεπτό για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Ε, η συγητής είναι ο Ντέρκ Φαν Έπινγκ, τον οποίο θα αντικαταστήσει ο κύριος Eugene Γιουτζίκα θα το ψηφίσουμε αύριο, οπότε ας είμαστε πολύ σύντομοι. Ε, στρέφουμε Αυτό το λέω και για τον εισηγητή και για τους κοινότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συναδέλφοι, το ECR είναι χαρούμενο που μετά από κάποιε διευκρινήσει ε, από αξιωματούχου τη ΕΣΜΑ ενημερωθήκαμε επαρκώ για του λογαριασμού, ώστε μπορούμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή για του λογαριασμού του 2018 για την Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, καθώ και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ένα άλλο ζήτημα, ωστόσο, είναι ο τρόπο με τον οποίο ο πρώην εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΑΤ ε, διορίστηκε ως ε, ανώτατο τέλεχος ε, της Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Αγορών στην Ευρώπη. Από το Φεβρουάριο του 2020 ο κύριος ε, Εμπιάν λέει ότι αυτή η, αυτό, η θέση δε, παρουσιάζει πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων. Αναφέρεται ότι αυτή η μεταπίδηση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να αποθαρρύνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ούτως ώστε να ε, επιβεβαιώνονται οι κατευθυντήρε γραμμέ της Κομισιόν του Διαμεσολαβήτρια και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κύριος εισηγητής λέει ότι τέτοια μεταπίδηση, ε, τέτοιε ε, υποθέσεις δίνουν ευκαιρία σε διάφορες ομάδες συμφερόντων να ανταμείβουν ρυθμιστέ για παρελθούσα συμπεριφορά και ανοίγουν την πόρτα για πιθανέ επιζήμιες ε, συμπεριφορές. Ε, ο εισηγητή του ECR θέλει να τονίσει ότι είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτή, διαφανή και ανεξάρτητη διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τι εποπτικέ ε, και τις λοιπές αρχές εντό τη Οικονομικής και Νομισματική Ένωση. Ο κ. Σεπίνγκ καλωσορίζει την πρόταση ψηφίσματο τη κυρία Τιλιάρη για τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών θεσεών. Οπότε υποστηρίζει το αίτημα προς το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΤ και το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΤ που επέτρεψε στον κύριο Φράκας να αναλάβει τη θέση CEO της ΑΦΜΑ και απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σχετικό πλαίσιο. Ο κύριος αναμένει μια επικοδομητική συνεργασία και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ που μου δώσετε και την ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ισκιώδης, ο κύριος Χριστοφόρου. Ε, θα πω ότι όσον αφορά την απαλλαγή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών της Χρηματοσυστατικής Εποπτείας που είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Θεωρούμε ότι και στι τρει γνωμοδοτήσει, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον ραπορτέρ, τον κύριο Νέπινγκ, ε, υπήρξαν οι αιτήσει λογαριασμοί για το 2018, είναι από κάθε πλευρά νόμιμε και κανονικέ. Θα υπερψηφίσουμε τη ε, πλειοψηφία των τροπολογιών, όμω υπάρχουν και ζητήματα για τα οποία έχουμε τι αμφιβολίε μα όσον αφορά την προσέγγιση τίθεται θέμα για την ανεξαρτησία των αρχών και ότι οι αρχέ δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητε όταν συνεισφέρουν τα κράτη. Αυτό όμω είναι ένα γενικότερο ζήτημα γιατί στο τέλο τη ημέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κατόπιν συνεισφορά των χωρών μελών. Δεν είναι μόνο για του εποπτικού οργανισμού, συνεισφέρουν οι χώρε μέλη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό και ολοκληρώνω γιατί γνωρίζω την πίεση του χρόνου που υφίσταστε ε, είναι όσον αφορά τα πλεονάσματα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι λογικό και δίκαιο να επιστρέφεται το 60% στις χώρες μέλη. Όμως τέτοιου είδες διευθετήσεις μπορούν να καταστούν εφικτές εάν και εφόσον υπάρξει διάλογο, δεν είναι δια τη επιβολή. Γι' αυτό και διαφωνούμε με την προσέγγιση ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή αυτή του καταμερισμού και να υπάρξει ένα επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την ανεξαρτησία των αρχών είμαστε αναφαντών υπέρ και για την αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό και υπερυποστηρίζουμε την ανεξαρτησία αυτών των οργανισμών και ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε διαφάνεια εφόλης της ύλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ζιλ από το Ρινιού. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ο δεν είναι εδώ. Οπότε έχω να αντικαταστήσει το Μόναρ. Παρακαλώ, γονάς, ζήτω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Μονάρ, δεν είναι εδώ, αλλά μου έστειλε κάτι για να σας το διαβάσω. Ο Μονά λέει λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι έχουν κεντρικό ρόλο αυτές οι ευρωπαϊκές αρχές στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθούν την σταθερότητα, την προστασία των καταναλωτών, είναι σημαντικές επίσης ε, στον τομέα της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης ε, και του ξέπλυματος μαύρου χρήματος και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πληρούν το καθήκοντά τους με τρόπο συνεκτικό, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό με επαρκείς πόρους και με ανοιχτή και ανεξάρτητη διοίκηση. Όμωνα ε, πιστεύει ότι οι περισσότερες τροπολογίες ε, θα ενισχύσουν το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή. Έτσι λοιπόν θέλει να σας ενθαρρύνει να ψηφίσετε υπέρ των τροπολογιών αυτών όπως προαναφέρθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα Ζήλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εισηγητή. Έχουμε ήδη συζητήσει το Δεκέμβριο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που έκτοτε λάβατε υπόψη πολλές ε, από τις ε, τροπολογίες που εμείς υποστηρίζουμε. Δείχνει ότι έχετε δείξει ανοιχτό πνεύμα και αυτό θα επιτρέψει να υιοθετηθεί αυτό το έγγραφο σε μια μορφή πιο ισορροπημένη, ε, με καλύτερες οι πιθανότητες να λάβει την πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβαστική τροπολογία όσον αφορά την ΕΜΕΦΑ. Είμαι και υπέρ της πρότασής σας ε, για προφορική τροπολογία όσον αφορά την γνωμοδότηση για την ΕΑΤ. Μεταξύ μας ε, παραμένει μία διαφωνία που έχει ήδη αναφερθεί όταν συζητήσαμε παλιότερα και που εξακολουθεί να υπάρχει για μας η έννοια της ε, σωστής επιστροφής, της σωστής συμβολή των κρατών μελών δεν είναι σαφής γιατί για μας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως το καταλαβαίνουμε δεν αντιστοιχεί σε αυτό και στη λίστα ε, ψηφοφοριών μας θα αντικατοπτρίζεται αυτή η θέση. Παρά τη διαφωνία σας ευχαριστώ για το σημαντικό σας έργο. Okay, thank you very much. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η διερμηνία σταματά εδώ, οπότε ε, στο εξή θα μιλήσουμε στα αγγλικά. Thank you.